Καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καταρχάς, πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη την οποία έχετε στους φακέλους σας. Αν δεν θέλει να πάρει κανείς το λόγο, αν δεν υπάρχουν, παρήνουμε την ημερήσια διάταξη δίχως τροποποίηση. Σημείο 2. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Να σας πω, καταρχάς, πρωτού ξεκινήσουμε τις εργασίες μας σήμερα το πρωί, ότι αύριο η Επιτροπή μας, η Ήτρε, θα συνεδριάσει στο 5G3, στην αίθουσα 5G3. Επομένως μην αφήσετε τα εγγραφά σας στην αίθουσα αυτή, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε την αίθουσα αυτή μόνο για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Δεύτερον, να σας πενθυμίσω ότι στις 2 Δεκεμβρίου, την επόμενη δηλαδή Δευτέρα, θα έχουμε εδώ στις Βρυξέλλες από τις 3 το μεσημέρι στις 6.30 μια συνεδρίαση στην αίθουσα Γιάν 2Q2. Πρόκειται για μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Βιομηχανίας όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια. Να σας πω επίσης ότι την επόμενη μετά Δευτέρα, την 9η δηλαδή Δεκεμβρίου, στο Στρασβούργο, θα διεξαχθεί μια συνεδρίαση από τις 7 ως τις 9 το βράδυ στην αίθουσα WIC 200. Πρόκειται για μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ας περάσουμε τώρα στην σημερινή ημερήσια διάταξη. Ξέρετε ότι έχουμε μια δημόσια ακρόαση σήμερα με θέμα την χρήση του αποθεματικού για νεοεισερχόμενους, δηλαδή του προγράμματος NER 300, καθώς επίσης και του σχεδίου ενεργειακής ανάκτησης για την ανανέωση του ενεργειακού τομέα. Καταρχάς προφανώς θα ήθελα να καλωσορίσω τους προσκεκλισμένους μας και εξ ονόματος της Επιτροπής μας να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας για την ακρόαση αυτή. Όσον αφορά τώρα την συνεδρίασή μας αυτή καθ' αυτή, να σας υπενθυμίσω ότι θα ολοκληρωθεί η δημόσια ακρόαση στις 11 ακριβώς. Επομένως, όλες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Ξέρετε ότι Πάντα θέλω να δίνω το λόγο σε όλους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να μοιράσουμε δίκαια το χρόνο που έχουμε στη θέση μας για την ακρόαση αυτή. Η ακρόαση χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα έχει να κάνει με το σχέδιο ανάκτησης ενέργειας και συγκεκριμένα με το πρόγραμμα NER300. Το δεύτερο τμήμα της δημόσιας ακρόασης έχει να κάνει με τις εμπειρίες που έχουμε μέχρι στιγμής με το πρόγραμμα NER300, ενώ το τρίτο τμήμα αναφέρεται στις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από το νέο αυτό πρόγραμμα. Ξεκινάμε ευθύ αμέσω, δίνοντας το λόγο για 10 λεπτά. Δυστυχώ ο πρώτος ομιλητής, ο κύριος Δελγκάντο Ρώσα, δεν έχει φτάσει ακόμα. Πρόκειται για τον εκπρόσωπο εκείνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα αναφερόταν στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης και ουσιαστικά στο πρώτο τμήμα της ημερήσιας διάταξης, καθότι λοιπόν απουσιάζει, μάλλον μόλις έφτασε. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει ευθύς αμέσως τώρα το λόγο ο κύριος Δελγκάτο Ρόζα. Μάλιστα, θα πάρει το λόγο λοιπόν όπως προβλεπόταν στην ημερήσια διάταξη. Έφτασε λοιπόν ο κύριος Σουμπέρτον Τελγκάντο Ρόζα και του δίνουμε ευθύ αμέσω το λόγο για 10 λεπτά. Thank you. My apologies for this delay. Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι που άργησα λιγάκι γιατί μπερδεύτηκα με, τα... με τις αίθουσες. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για το θέμα μου παρόλο που μόλις μπήκα. Και θέλω να σας ενημερώσω λίγο για αυτό το ε, πρόγραμμα το οποίο, για το οποίο μόλις ακούσατε και για το πώς θα μπορέσει να ανανεώσει τον ενεργειακό τομέα. Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ε, και και βεβαίως ε, εργάστηκα και εγώ στην εκπόνηση αυτού του προγράμματος. Ε, NER 300. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν ε, δίνει οικονομική ενίσχυση σε λίαν καινοτομικά προγράμματα ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης άνθρακος, δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακος η, ονομασία του NER 300 προέρχεται επειδή ακριβώς καλύπτει 300 εκατομμύρια ε, ευρώ για τις ενισχύσεις και κάναμε τον πρώτο γύρο της νομισματοποίησης ε, διαθέτοντας 200 εκατομμύρια ε, τα οποία τελικά αυξήθηκαν σε 300 και για συνολική χρηματοδότηση 1,5 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για τον όλο τομέα. Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Δέσμευσης, ε, ανάκαμψης, Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης, Επίσης ε, καλύπτει τη χρηματοδότηση αιωλικής ενέργειας και προγραμμάτων δέσμευσης και αποθήκευσης. Το budget είναι 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 0,6 θα χρησιμοποιηθούν για υπεράκτιες ε, ενεργειακά αιωλικά πάρκα και 1 δισεκατομμύριο για προγράμματα δέσμευσης και αποθήκευσης. με όλα, αυτά τα προγράμματα και ενισχύσει, στόχος μας είναι να η ενεργειακή ε, διαφοροποίηση ε, όσον αφορά την παροχή ενέργειας και να ολοκληρώσουμε ομαλά την εσωτερική ενεργειακή αγορά μειώνοντας τα αέρια του θερμοκηπίου. Τώρα, πώς συνδέεται το NER300 με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκτησης, το EEPR και τα δύο συγχρηματοδοτούν ε, υπεράκτια αεολικά πάρκα και προγράμματα δέσμευσης και αποθήκευσης και επίσης προσφέρουν χρηματοδοτική ενίσχυση σε όλων τους τύπους της ανανεώσιμες ενέργειας. Το NER 300 <clears throat> θα πρέπει η χρηματοδότησή του να μειώνεται όταν λαμβάνει ενισχύσεις από το EEPR. Τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα του NR300 μετά την πρώτη δημοσιοποίηση των ε, μειοδοτικών ε, για, πρόσκληση, ε, για υποβολή αιτήσεων, για χρηματοδότηση προγραμμάτων. Το Δεκέμβριο 2012 η Κομισιόν διέθεσε περισσότερο από 1,2 δισεκατομμύρια σε 23 λίαν καινοτομικά προγράμματα νεώσιμης ενέργειας. Ε, Παραδείγματο χάρη, βιοενέργεια, προηγμένα βιοκάψιμα, συγκεντρωτική ηλιακή ενεργειακή ισχύ, γεωθερμική ενεργειακή ισχύ, ε, αιωλική ενέργεια, ενέργεια από του ωκεανού και έξυπνα δίκτυα. Και ε, με αυτά τα χρήματα, με αυτή τη χρηματοδότηση εντάξαμε 16 κράτη-μέλη. Και βεβαίως όλη αυτή η χρηματοδότηση βασίστηκε στα κριτήρια επιλεξιμότητας, ε, τα οποία ε, κριτήρια περιλάμβαναν και νοτομική τεχνολογία και τη δυνατότητα αύξησης και διεύρυνση του προγράμματος προγράμματα αυτά θα, η τελική τους χρηματοδότηση θα αποφασιστεί προς το τέλος του 2014 και θα ισχύσουν μέχρι το 2016 που θα είναι και η τελική ημερομηνία για να ξεκινήσει η λειτουργία τους. Τώρα, πώς, με ποια κριτήρια διατίθεται η χρηματοδότηση για προγράμματα δέσμευσης και αποθήκευσης. Υπάρχουν ε, πολλές, ε, πολλά αίτια για τα οποία υπάρχουν χρηματοδοτικά κενά. Ή τα προγράμματα δεν είχαν προχωρήσει αρκετά ή το χρονικό διάγραμμα δεν ήταν σωστό ε, στην πρώτη πρόσκληση υποβολή αιτήσεων. Αλλά μέχρι τώρα ένα κράτος μέλος έχει υποβάλει ένα πρόγραμμα CCS, δέσμευσης και αποθήκευσης και συνεχίζεται η διαδικασία εξέταση μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Τώρα πώς θα υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως όσον αφορά την ανάκτηση, διότι όταν χρειάζεται ανάκτηση τα οικονομικά στοιχεία υπερισχύουν. Όμως υπάρχει και μία, μία ανάγκη της αγοράς παροχής ενέργειας σε χαμηλότερη τιμή και γι' αυτό πρέπει να πιέσουμε πολύ ε, έντονα την ε, ε, ενσωμάτωση καινοτομικών προγραμμάτων. Επίσης, εάν δεν εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα, τότε θα έχουμε και πολύ λιγότερα έσοδα από τα προγράμματα CCS, δέσμευσης και αποθήκευσης. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεπεράσουμε την χιονοστιβάδα των κριτηρίων τα οποία έχουμε, με των περιθωρίων που έχουμε και να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά προγράμματα. Στην κλιματική διάσκεψη που έγινε στη Βαρσοβία, συζητήσαμε βεβαίως και σχολιάστηκε το μήνυμα για το, για το κλίμα, για την ατμόσφαιρα και όλα τα συναφή προβλήματα, παραδείγματο χάρη τα ορυκτά καύσιμα και η υπερβολική εξάρτηση από αυτά και η χρήση τους. Πρέπει λοιπόν ακριβώς ε, να ε, διαδώσουμε αυτό το μήνυμα και να πούμε ότι μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί ε, και να, να ολοκληρώσουμε καλύτερα, με, με, με βέλτιστα όλα αυτά τα προγράμματα δέσμευσης και αποθήκευσης. Αλλά βλέπετε ότι εδώ εμπλέκονται και δημόσια κονδύλια. Όχι μόνο για τα προγράμματα CCS, αλλά και για πολλά άλλα προγράμματα, παραδείγματο χάρη και για την βιομηχανία τις εκπομπές καυσέριων. Δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις οι οποίες πιέζουν, αλλά υπάρχουν και τα θέματα των ε, αγωγών παραδείγματο χάρη των, και των λόμπις, των ομάδων πιέσεων. Και πολλές φορές υπάρχει μία διαμάχη μεταξύ συμφερόντων, η οποία φάνηκε ε, στην διάσκεψη για το κλίμα. Εάν, λοιπόν, το NER 300 ε, δεν δεν έχει προβληθεί πολύ. Είναι γεγονός όμως ότι υπάρχει, υπάρχουν έντονα επιχειρήματα που το υποστηρίζουν και ιδίω από την πλευρά της αγοράς και των επιχειρήσεων. Είχα μία σχετική εμπειρία Δηλαδή το πρώτο ε, πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε στην Ιταλία από το NER 300 ήταν το πρόγραμμα το λεγόμενο BEST, το οποίο ε, ξεκίνησε το 2013 και είναι πρόγραμμα βιοενέργειας δεύτερης γενιάς. 28 εκατομμύρια ευρώ έλαβε και ο στόχος ήταν να μετατρέψει την ε, λιγνοκυταρική βιομάζα χαμηλής ποιότητος σε υψηλής ποιότητος εθανόλη. Το πρόγραμμα ε, αναπτύχθηκε ε, σε εμπορική κλίμακα για την χρήση κυταριού εθανόλη στον κόσμο, διεθνώς. Δηλαδή, μετατρέπουμε ε, μία χαμηλή βιομάζα, χαμηλής ποιότητας σε υψηλής ποιότητας εθανόλη και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα. Το δεύτερο, η δεύτερη εμπειρία που είχα, που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό να λειτουργεί το 2014, στην αρχή του 2014, ε, είναι το δεύτερο πρόγραμμα NER 300, είναι το γερμανικό Verbio Δηλαδή ένα πρόγραμμα στην περιοχή του Ούκερμαρκ στην Γερμανία το οποίο θα δημιουργήσει αέρια με αναεροβική ζύμωση και θα χρησιμοποιήσει 70.000 τόνους άχυρο και θα χρηματοδοτηθεί με 22 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, τι έχει προσφέρει το πρόγραμμα NR300 e για την καινοτομία, την πράσινη ανάπτυξη και την απασχόληση. Μέχρι τώρα τα προγράμματα αυτά ε, θα ε, εκμεταλλευτούν την υπάρχουσα εμπειρία και την αλυσίδα καινοτομιών και θα προσπαθήσουν το πρόγραμμα αυτό να ξεπεράσει τα βασικά εμπόδια και προσκόμματα στην ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας τεχνολογιών. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους, ε, στο ξεπέρασμα εμποδίων και Μέχρι τώρα το πρόγραμμα έχει δώσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσει ε, το οποίο ε, συμπληρώθηκε με 2 δισεκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικές επενδύσεις. Μιλάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή για 3,2 συνολική χρηματοδότηση, 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πολύ μεγάλος αριθμός διότι ε, συνάδει και με την ενίσχυση της αγοράς ε, εργασίας. Ε, τώρα, βράχει πρόθεσμα θα προσθέσουμε 100 τετραβατόρες στην ενεργειακή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό βεβαίως ισοδυναμεί με τα κάρτα προς χρησιμοποιούν ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα το ετησίως αλλά το 1.300 300 e θα βελτιώσει και την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο ε, και θα ε, αποδειχθεί πολύ ανταγωνιστικό. Έχουμε και άλλα ε, και, καινοτομικά προγράμματα τα οποία θα καλυφθούν από το 1.300 300 e με βάση την, το, το στόχο δέσμευσης και αποθήκευσης. Πιστεύω ότι το NER300 <clears throat> θα πρέπει να συνεχιστεί να έχει ένα follow-up ε, δεδομένου ότι η δεύτερη πρόσκληση για υποβολή ε, αιτήσεων ε, ξεκίνησε τον Απρίλιο 2013 και η επιλογή των προγραμμάτων που θα καλυφθούν ακόμα συνεχίζεται και η δεύτερη και θα αποφασιστούν τον Ιούνιο του 2014 ποια θα χρηματοδοτηθούν. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Τελγκάτο Ρόζα. Έχουμε στη θέση μας 20 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο κύριος Κανσάν είναι πρώτος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω κύριε Ντελγκάντο Ρόζα για την παρουσίασή σας. Μία συγκεκριμένη ερώτηση θέλω να κάνω. Μιλάμε πάρα πολύ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολύ σωστά το κάνουμε βέβαια αυτό. Αλλά όταν τελικά συνδέουμε με το δίκτυο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες τις δυνατότητες που μας δίνουν, τότε ξέρουμε ότι το τμήμα εκείνο της ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται το πετάμε τελικά, δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Επομένως, το όλο ζήτημα της αποθήκευσης της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να αποθηκεύουμε την ενέργεια αυτή και να τη χρησιμοποιούμε όταν την έχουμε ανάγκη. Ξέρετε ότι καταλήγουμε τελικά πολύ συχνά να έχουμε πλεονάζουσα ενεργεία, την οποία όμως δεν χρησιμοποιούμε. Επομένως, το ερώτημά μου είναι το ακόλουθο. Η όλη αυτή η εργασία που λαμβάνει η χώρα και που έχει να κάνει με την αποθήκευση της ενέργειας, τη συγκέντρωση και την αποθήκευση της ενέργειας, προκειμένου αυτή να μην πηγαίνει χαμένη στη συνέχεια. Πώς μπορεί να μας δώσει κάποιες λύσεις σήμερα, πώς μπορούμε να επιλύσουμε μέσω της αποθήκευσης το πρόβλημα αυτό της μη χρησιμοποίησης τελικά της ενέργειας. Ακούσαμε διάφορες προτάσεις, αλλά δεν μπορώ εγώ να καταλάβω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, τι ανάλυση έχει γίνει για το ζήτημα αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα αυτό και θεωρώ ότι είναι απόλυτα λογικό να καταλήξουμε σε μια σωστή λύση η οποία θα καταφέρει να μας βοηθήσει για την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας. Σας ευχαριστούμε κύριε Κανσιάνο, κύριος Πρόντι, το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι το CCS, η αποθήκευση δηλαδή και η... η δέσμευση άνθρακα μπορεί να είναι η τέλεια λύση. Και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον άνθρακα όπως το κάναμε ως τώρα ή όπως το υπολογίζαμε. Επίσης πρέπει να γίνει σαφές ότι το σύστημα στόχο θα πρέπει να έχει να χρησιμοποιεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και να αξιοποιεί την αποθήκευση, το storage, με συστήματα που δεν χρησιμοποιούν την καύση, αλλά την μετατροπή των βιοκαυσίμων και των ορυκτών καυσίμων, καθώς και της βιομάζας, και μπορούν να τα μετατρέπουν όλα αυτά σε αέριο. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιείται οξυγόνο ή ατμός και δεν θα υπάρχει πρόβλημα διαχωρισμού του διοξιδίου του άνθρακα από άλλα αέρια τα οποία δεν θέλουμε στην ε, καύση όπως το άζωτο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι να δούμε εάν μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συστήματα ε, ή όχι. Εγώ δεν νομίζω ότι με τη συμβατική καύση μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το σύστημα, τουλάχιστον όπως μας έχει παρουσιαστεί ως τώρα. Πιστεύω επίσης ότι το πρόβλημα που τίθεται είναι ακριβώς να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενέργεια. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρξει δίκτυο με μεγάλες ικανότητες μεταφοράς, όπως ε, συνεχούς υψηλής τάσεως. Ένα δίκτυο που να συνδυάζει την χρήση ελληνικής ενέργειας και της ε, υδροηλεκτρικής Δηλαδή, να μπορούμε να έχουμε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να έχουμε ως στόχο. Έπειτα, ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες αποθήκευσης. Μπορεί με την παραγωγή υδρογόνου ή με τις αντλίες να πετύχουμε κάτι ή η ενέργεια η είναι ήδη μια μορφή παροχής ενέργειας. Ευχαριστούμε ο κύριος Δέβης. Ευχαριστώ. Σημάμαι τις τροπολογίες για το NER 300 το 2008 και ήμουν εισηγητής τότε για το πρόγραμμα CCS, δέσμευσης και αποθήκευσης. Ε, με συγχωρείτε λοιπόν που θα επανέλθω στο ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης. Ο David Hown, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής του τμήματος κλίματος στη Shell και αυτός είχε την ιδέα και μαζί με την κυρία Doyle Είχαμε τότε συζητήσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο το 2008 για να βρούμε ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στην πρακτική της ε, δεσμεύσης ε, για την αποθήκευση, μείωση διεξιδίου του άνθρακος κλπ. μέχρι το 2015. Υπέγραψαν τις ε, δεσμεύσεις για θεωρητικά δηλαδή για όλα αυτά τα ωραία πράγματα αλλά δεν είχαν αποφασίσει από πού θα προέλθουν τα κονδύλια. Σε 600 εκατομμύρια ήταν τότε το ποσό του NER όταν είχα υποβάλει τότε την πρώτη τροπολογία και μειώθηκε στο ε, ε, πρώτα μειώθηκε στα 500 μετά έχουμε ένα μεγάλο καυγά με το συμβόλιο. Ε, συμβούλιο μετά έγινε 300. Ε, βεβαίως τότε είχαμε δυσκολίες να πείσουμε τον κόσμο αλλά χαιρόμεθα ιδιαίτερα που βλέπω ότι τώρα έχουν πιστεί πολλά στελέχη και εγώ το αποκαλώ πάντοτε n NER, όχι NER, όπως λένε μερικοί. Τώρα, πού βρισκόμαστε σήμερα. Τρία στοιχεία. Πρώτα, έχει διασυνδεθεί με το πρόγραμμα δέσμευσης και αποθήκευσης και τις καινοτομίες. Ε, υπάρχει λοιπόν μία διασύνδεση. Πρέπει ε, λοιπόν να επανέλθουμε στην έμφαση που δίνεται στη δέσμευση και αποθήκευση. Εκεί ήταν το επίκεντρο, ο στόχος μας. Τώρα πόσο, πόσα από εσά θα πάνε στις ανανεώσιμες. Ε, ε, ενεργειακά δηλαδή, στα ανανεώσιμα. Ε, και είχαν, είχε πει τότε ο Επίτροπος ότι όχι πάνω από 60% ε, θα πάνε στα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά τελικά όλα τα κονδύλια πήγαν για τα ανανεώσιμα και αυτό, αυτό δεν ήταν ο στόχος μας διόλου στην αρχή. Και τελικά κατέρευσε η τιμή ε, του άνθρακα ενώ είχαμε πει ότι θα ε, μαζέψουμε 9 δισεκατομμύρια ευρώ τελικά μαζέψαμε 6 ε, δις και αυτή τη στιγμή το πολύ να, να μαζέψουμε 2-2,5 δισεκατομμύρια διότι έχει συντριβήσει θλιβή η τιμή του άνθρακα η, το, το Δεκέμβριο του 2008 υιοθέτησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το πρόγραμμα NER 300. Και τέσσερα χρόνια μετά από αυτό, τέσσερα χρόνια χρειάστηκαν για να διαμορφωθεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο ε, με ανανεώσιμα, καινοτομίε κλπ. Αυτό είναι υπερβολικά αργά, άργησε υπερβολικά πολύ όταν η Κίνα σε μπορούμε να πούμε ε, ταχύτατο χρόνο, σε χρόνο μηδέν ξεκινάει τέτοια προγράμματα και βρίσκει και τη χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε ε, έντονα. Ε, το, το δεύτερο στοιχείο είναι η ευελιξία του μηχανισμού. Ένας από τους λόγους που αργήσαμε τόσο πολύ να υλοποιήσουμε το, το, το σύστημα είναι επειδή μας πήρε πολύ χρόνος να σχεδιάσουμε τους κανόνες. Είναι αρκετ, θα έλεγα, δεν έχει την ευελιξία που χρειάζεται ε, και θα πρέπει να τις εισαγάγουμε. Ε, πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα, τι ενισχύσεις θα χρειαστούν και ποια υπουργεία, δηλαδή ποια δημόσια διοίκηση, ας πούμε το Υπουργείο Οικονομικών, θα δώσει τις εγγυήσεις ε, χρηματοδότησης για να προστατευθεί η ε, χρηματοδότησή τους, τα δάνεια κλπ. Πρέπει λοιπόν να ακούσουμε και τον ιδιωτικό τομέα και να εξασφαλίσουμε την καλύτερη χρήση των δημοσίων κονδυλίων. Ξέρω ότι πολλοί στην Κομισιόν υποστηρίζουν ένα νέο καινοτομικό ταμείο για να ενισχυθούν τα προγράμματα CCS. Εάν λοιπόν υπάρξει ένα νέο μήνα ε, πηγή χρηματοδότηση για τα ECCS θα πρέπει αυτό να, είναι, να γίνει, να εδρεωθεί ταχύτερα, καλύτερα και με τα απαραίτητα κονδύλια. Η Πρόεδρος. Ο κύριος Ντέιβις έχει περισσότερο χρόνο γιατί είναι εισηγητής στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Τώρα ο λόγος στην συνάδελφο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Okay. το πρόγραμμα. Είναι πολύ θετικό και ελπίζαμε ότι θα δημιουργήσει προσδεθεμένη αξία. Όμως από ακούσαμε και από τον συνάδελφο, είναι ανησυχητικά τα νέα. Έξι προγράμματα CCS ξεκίνησαν από το 2008 και τώρα δεν ξέρουμε τι θα απογίνει. Έχουμε ένα παράδειγμα από το Ενωμένο Βασίλειο. Και αυτό αρκεί. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξή. Ξέρω ότι ένα ε, πρόγραμμα θελοποιείται και στην ε, ε, Πολωνία, στο Ντουργκάντοφ, στο εργοστάσιο παραγωγής, μικτής παραγωγής εκεί. Τι θα κάνουμε με το θέμα αυτό, γιατί κάποιοι λένε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι αρκετά ασφαλής. Βασίζεται στην αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα σε παλιά ορυχεία. Ότι αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο ιδίω ορισμένε περιοχέ. Έχω διαβάσει σχετικά δημοσιεύματα και άρθρα. Ανησυχεί ο κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω αν αυτό αληθεύει. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τελικά δεν υλοποιήθηκαν λόγω της ε, θέσης των εργοστασίων παραγωγής κοντά σε αστικά κέντρα. Επίσης κάτι άλλο που λέγεται σε πολλά άρθρα είναι το κατά πόσον κατά πόσον ε, υπάρχει κίνδυνος από αυτού του είδους την ε, μέθοδο. Ακούγεται παράλογο, ίσως να είναι υπερβολικό, αλλά κυκλοφορεί πολύ αυτό και υπάρχουν σχετικές έρευνες, το ξέρω, αλλά θα ήθελα να ξέρω πόσο έχει προχωρήσει η έρευνα. Ε, σε τι βαθμό ξέρουμε το κατά πόσον είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται το, το άνθρακα στην χημική βιομηχανία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή βιώσιμε μέθοδοι για την χημική βιομηχανία. Ήθελα να δοθεί έμφαση σε αυτό αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χέρτσοκ. Thank you. Uh, thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Ντελγκάδο, ελπίζαμε η Επιτροπή να μας εξηγήσει καλύτερα την ε, αξία του NER. Μέχρι το 2008 για το ε, NER το 300 θεωρούσαμε ότι η χρηματοδοτική στήριξη είναι απαραίτητη για να υλοποιηθούν σχετικές πολιτικές. Ήθελα όμως να μας πείτε κι εσείς πού βλέπετε την υποστηθέμενη αξία ακριβώ στα προγράμματα αυτά. Βλέπετε να υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση ε, και πιστεύουμε ότι μεγάλο μέρος της δέσμευσης που βλεπετε την υποστηθεμενη αξια ακριβως στα προγραμματα αυτα χαθεί οφείλεται στην, ε, στις καθυστερήσεις. Πού είναι αυτή η προστεθέμενη αξία που περιμέναμε. Είναι πολλές οι κριτικές από πολλούς τους συναδέλφους διότι πολλά από τα προγράμματα CCS δεν έχουν προχωρήσει όπως περιμέναμε και κάνουν μεγάλη προσπάθεια οι συνάδελφοι για να πείσουν τους υπόλοιπους ότι έχει νόημα το όλο αυτό εγχείρημα. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το διοξείδιο του άνθρακα, χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες εξηγήσει. Πού βλέπετε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και εάν δεν τη βλέπετε, πού χάθηκε και τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Εάν δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει, να δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Δελγκάδο Ρόζα για να τον παρακαλέσω να απαντήσει στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις, ακόμη και τις κριτικές που ακούστηκαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και για λόγους χρόνου. Πρώτο θέμα, η αποθήκευση και τι γίνεται με την ανανεώσιμη ενέργεια όταν δεν είναι πάντα του διαθέσιμη εφόσον τη χρειαζόμαστε. Αυτό είναι ένα σαφώ ένα θέμα, το οποίο όμω μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν θέλετε να δούμε τι γίνεται στο πολύ μακροπρόθεσμο μέλλον, στο τέλο, η βιώσιμη ενέργεια θα είναι ανανεώσιμη σε κάθε περίπτωση, ασχέτω του πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Υπάρχουν ευτυχώ πολλέ πηγέ ανανεώσιμη ενέργεια και κάποιε από αυτέ είναι και αλληλοσυμπληρωματικέ. Εάν σκεφτείτε δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια σε συνδυασμό με την πράσινη ενέργεια, το πώ η, η ενέργεια από το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω υδραυλική ενέργεια για την αποθήκευση, ε, αυτά μπορούν να συνδυαστούν και με τη νύχτα ή την διαθεσιμότητα ηλιακή ενέργεια Βεβαίω, για να ολοκληρωθούν όλα αυτά χρειαζόνται τα ευφυή δίκτυα για να μας επιτρέψουν να αντλήσουμε από εκεί που θέλουμε την ενέργεια και να την πάμε ε, στο σημείο που θέλουμε επίσης. Είμαστε σε ένα στάδιο όπου δεν μπορούμε βεβαίως από τα ορυκτά καύσιμα με μια κίνηση να αντλήσουμε αυτό που θέλουμε. Είναι ακόμη ένα πρόβλημα, γιατί έχουμε ακόμα μεγάλη ανάγκη από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται. Τώρα, συνολικά, εάν ε, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα είναι σωστή προσέγγιση, ε, εάν θέλετε να παραμένει ο άνθρακα όσοι έχει και να μην χρησιμοποιηθεί, Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά αν παραμείνουμε στην καύση, πάλι θα υπάρχει απώλεια ενέργειας. Ε, εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται σε μια μεταβατική περίοδο όπου ακόμη έχουμε κάποια εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν χρειαζόμαστε βεβαίω όλα τα ορυκτά καύσιμα, αλλά αυτά που χρησιμοποιούμε δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι και όλο ο άνθρακα που εκλείουν να διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα. Πρέπει ο άνθρακα να επιστρέφει στην γη, εκεί όπου ανήκει. Το CCS από όλε τι ερευνέ μα έχει προκύψει ότι είναι απολύτω ε, αναγκαίο μέθοδο. Τι γίνεται με τη βιομάζα τώρα και το CCS. Εδώ τι χρειάζεται να γίνει από το διοξίδιο του άνθρακα και την γη ε, και το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει συμπληρωματικότητα. Τώρα, για τα υπερδίκτυα, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό πρόβλημα είναι να προχωρήσουμε με διαφορετικούς δρόμους. Όχι μόνο με το CCS ή μόνο με τα ευθύ ή μόνο με τον συνδυασμό τώρα για τα σχόλια του ε, κυρίου Ντέιβις για το ΝΕΡ 300. Ε, Όσοι βλέπουν το πρόγραμμα αυτό σε ένα πρόγραμμα CCS και μόνον δεν θα είναι ικανοποιημένοι. Δεν είναι απόλυτη επιτυχία του, αλλά σε ό,τι αφορά την προστιθεμένη αξία. Τότε δεν ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω τι ενθουσιασμό είχε τότε η Επιτροπή ή όχι. Όμως αν το δούμε από κυβερνητική σκοπιά, η συζήτηση δεν είχε στόχο το CCS να καλύπτεται μόνο από το NER. Ε, κάποιοι ε, αντιτίθεντο στο CCS και κάποιοι θέλαν να είναι δίπτυχο και να αφορά μόνο τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Τώρα, εάν το πρόγραμμα έχει πλαισιώσει μόνο το CCS και τι υψηλά ανανεώσιμε, υψηλή υψηλής, ε, ανανέωση πηγέ ενέργεια, τότε Ήδη έχετε την απάντησή σας για την προστιθέμενη, ε, για την προστιθέμενη αξία. Το εργοστάσιο που σας ανέφερα στο Πιεμόντε είναι από εμπορική πλευρά τελείως βιώσιμο. Δηλαδή παίρνουμε την ενέργεια που θέλουμε από την πηγή που θέλουμε και την πηγαίνουμε στο σημείο που θέλουμε. Θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλά τέτοια εργοστάσια στην Ευρώπη και επίσης εκτός Ευρώπης με ευρωπαϊκή τεχνολογία. Είναι πολλές τέτοιες εργασίες που μπορούμε να δημιουργήσουμε και αντλούμε και περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια, μειώνουμε τι εκπομπέ και ε, καλλιεργούμε τι ανανεώσιμε πηγέ. Υπάρχει λοιπόν αρκετή προστιθέμενη αξία τη δική μας την πλευρά. Ε, ναι, υπάρχει προστιθέμενη αξία με το CCS. Τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση του ενός ή του άλλου προγράμματος από την πλευρά του λόγου χάρη, του τι έγινε στην Πολωνία λόγου χάρη. Ναι, υπήρχε ένα πρόγραμμα που ήταν ε, υποψήφιο και για το EPR και για το NER300. Όμως έχουμε 10 βιώσιμα προγράμματα CCS και σε πρώτη φάση ένα προς ένα μερικά εγκαταλείφθηκαν. Ο πιο σημαντικός λόγος ήταν συνήθως ε, η έλλειψη χρηματοδότησης. Τώρα στον Μπέρτσακοφ, όπως είπατε κι εσείς, υπήρξε ένα πρόβλημα χρηματοδότησης πολύ σοβαρό και άλλες πτυχές προβληματικές, όπως η τεχνική αβεβαιότητα ή ότι η οδηγία CCS δεν είχε ακόμη υλοποιηθεί, μεταφερθεί μάλλον στην Πολωνία σε αυτή την περίπτωση και θέματα αποδοχής από το κοινό, από το, τους πολίτες. Η πρόσληψη δηλαδή της κοινή γνώμης δεν αρέσει σε όλους η δέσμευση άνθρακα και η αποθήκευσή της στη, στη γη. Όμως η οδηγία CCS, το πώς θα παρουσιαστεί, ε, και πώ θα υλοποιηθεί ακριβώ στην πράξη είναι ένα θέμα που εξαρτάται από εμά. Το θέμα τη πρόσληψη από το κοινό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εάν θέλουμε να είναι βιώσιμη λύση το CCS. Σε ορισμένε περιπτώσει για του Ευρωπαίου δεν υπάρχει πρόβλημα, σε κάποιου ε, όμω φαίνεται κάτι τελείω αδιανόητο. Δεν του φαίνεται ασφαλέ να αποθηκεύεται άνθρακα εκεί που μπορεί να υπήρχε ένα ορυχείο ή που μπορεί να υπήρχαν ε, υδροφόροι ορίζοντε ή οτιδήποτε άλλο. Η ε, στάση λοιπόν της κοινή γνώμη είναι ένα θέμα. Η ασφάλεια δεν είναι πρόβλημα από τη δική μας την Σκοπιά, αρκεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Τώρα, υπάρχουν κάποιες βιομηχανικές χρήσεις όπου το διοξίδιο του άνθρακα μπορεί να αξιοποιηθεί και εκεί προκύπτει όφελος. Το θέμα είναι όμως πώς εμπορικά θα το αναπτύξουμε αυτό και αν από, ποσότητας, από την πλευρά της ποσότητας έχει ενδιαφέρον. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε με μεγαλύτερη προσοχή την αποθήκευση του άνθρακα και τη χρήση. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντελγκάντο Ρόζα για τις απαντήσεις αυτές που δώσατε, ανταποκρινόμενος στις διάφορες παρατηρήσεις που γίνανε από τους συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και συνεχίζουμε τις εργασίες μας με τρεις παρουσιάσεις, οι οποίες θα γίνουν η μία μετά την άλλη. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα της δημόσιας ακρόασης, εμπειρίες από την χρήση του προγράμματος NER300. Πρώτος θα πάρει το λόγο ο κύριος Ζάκα Κιβιέτε, όσον αφορά τις προοπτικές πρόγραμμα του, στα πλαίσια του προγράμματος Νέα 300, καθώς επίσης και τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει. Καλημέρα σε όλους. Και είμαι εκπρόσωπος της Early Kid. Είμαι Business Control Manager. Και ασχολούμαι ιδίως ε, κυρίως με τα προγράμματα δέσμευσης και αποθήκευσης CCS στο Rotterdam της Ολλανδίας. Έχω τέσσερις διαφάνειες που παρουσιάζουν το περίγραμμα και την ουσία του προγράμματος και την εμπειρία μας ε, στο NER 300 και γιατί αποτύχαμε και τις δυσκολίες ανάπτυξης του CCS για τη βιομηχανία. Okay. you see here... Καταρχάς βλέπετε εδώ μία εικόνα της Air Liquide. Είμαστε μία πολύ μεγάλη ε, βιομηχανία παροχής ε, We deliver here oxygen, nitrogen. Υγραερίου. Υγρού φυσικού αερίου, υγραερίου. Και βλέπετε την κόκκινη, τον κόκκινο αγωγό ε, είναι η παροχή υδρογόνου και η κόκκινη είναι η παροχή ε, αζότου, αζότου και οξυγόνου. Βλέπετε τις, ε, τους τρεις χρωματισμούς. Και έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο δίκτυο διανομής υδρογόνου, τεράστιο δίκτυο και είχαμε προτείνει να ανακτήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα στις εγκαταστάσεις μας στο Ρότερνταμ ε, και εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα των έργων, των projects. Το χάρτη, το χάρτη, τον οδικό χάρτη το, μεταφορών δικών μας, δηλαδή του Ρότερντα, εδώ ε, το πορτοκαλί είναι η ανάκτηση διοξιδίου του άνθρακος ε, από πηγές στο λιμάνι του Άμστερνταμ και εν συνεχεία διανομή του σε πράσινα προγράμματα. Βλέπετε τον αγωγό, το πράσινο, το ανακτημένο δηλαδή, ε, το οποίο ιδίω το καλοκαίρι καθαρίζεται και εκλείεται στον αέρα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται ε, ένα πρόγραμμα DDF το οποίο ανακτά το διοξείδιο του άνθρακο από, από μια εγκατάσταση καύσης άνθρακα. Το πρόγραμμά μας είχε το στόχο από, ένα, από μια εγκατάσταση υδρογόνου να ανακτήσουμε το διοξίδιο του άνθρακο. Είναι δικό μας πρόγραμμα της εταιρείας της Αρλικίδ και μετά θα συνεργαζόμασταν σε ένα κονσόρτσιο με το λιμάνι του Ρότερνταμ και ε, θα ε, παρέκλεινε ο αγωγός προς την περιοχή μας φλάκτα όπου θα συνδεόμασταν με τα ευρωπαϊκά προγράμματα έστε ώστε να μοιράσουμε το κόστος και καλύτερες, να είχαμε και καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και στη δεύτερη φάση είχαμε την πρόθεση μέσω ενός σταθμού ε, διοξιδίου του άνθρακα να μπούμε και στα πετρελαϊκά ε, χωράφια, αν θέλετε. Διότι πιστεύουμε ότι αν καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τον εκτιμένο διευθύνιο του άνθρωπο, προσφέρουμε θέμενη αξία και δεν δημιουργείται πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα, αλλά λαμβάνει και κάποια αξία. Ε, βλέπετε λοιπόν εδώ την συνέργεια μεταξύ αποθήκευσης και μεταφοράς, διότι σαφώς ε, χρειάζονται συνέργειες διαφορετικά. Είναι υπερβολικό το κόστος και ε, θα είχαμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε και το ε, ανακτημένο διοξίδιο του άνθρακα. Συνεργαστήκαμε με πολλές εταιρείες, όλες οι εταιρείες συνέβαλαν με τις εμπειρογνωμοσύνες τους και τις τεχνολογίες τους. το χάρη το λιμάνι του Ρότερνταμ είχε την υποδομή. Είχαμε ε, ναυτιλιακή εταιρεία η οποία μεταφέρει ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Όλοι λοιπόν είχαν την, ε, είχαν την εμπειρογνωμοσύνη τους που χρησιμοποίησαν σε αυτή τη συνέργεια και είχαμε καλή υποστήριξη από τις τοπικές αρχές, από την κοινότητα του Ρότερνταμ, από το λιμάνι του Ρότερνταμ. Ε, και αυτή ήταν η βάση του προγράμματός μας. διαθέσαμε τέσσερα χρόνια για ε, διαθέτοντας τη χρηματοδότηση για, την, για αναπτυξιακά έργα και για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του προγράμματος. Από οικονομικής πλευράς είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι με αυτά τα, τις τιμές του ETS δεν κερδίζουμε χρήματα. Έπρεπε όμως να το χρηματοδοτήσουμε, διότι ε, χρησιμοποίησαμε την ίδια αποθήκευση και την ίδια αποδομή με την οδική αποθήκευση. Δεν είχαμε ευτυχώς ε, ε, προβλήματα αποδοχής από το, τους πολίτες, δηλαδή την, από τις κοινότητες και χρησιμοποίησαμε και μία δημόσια επιδότηση και ε, στείλαμε και μια επιστολή στο ε, Ολλανδικό κράτος που επιβεβαιώσαμε, επιβεβαιώσαμε την πρόθεσή μας για το έργο. Αλλά για το NER 300 είχαμε μία αίτηση από την κυβέρνηση να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία. Και τα οικονομικά στοιχεία που μας ήρθαν από την πλευρά της κυβέρνησης δεν ήταν ταυτόσιμα με τα δικά μας είπαμε ότι για λόγους ανταγωνιστικότητος και εμπιστευτικότητος δεν μπορούσαμε εμείς να αποκαλύψουμε τα οικονομικά μας στοιχεία και γι' αυτό κολλήσαμε και κόλλησε και όλο το έργο. Είχαμε αργότερα μία συνεδρίαση για να ε, εξηγήσουμε, να διευκρινίσουμε ορισμένες θέσεις μας και να ε, προβάλλουμε τη στάση μας, ε, την προσέγγιση μας, αλλά δεν υπήρχε συμφωνία, δεν υπήρχε σύμπτωση απόψεων. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Δεν δέχτηκαν τις εξηγήσει μας, ήταν πολύ αργά, δεν υπήρχε, όπως είπα, συμφωνία μεταξύ ε, του Δημοσίου και ημών και έτσι σταμάτησε το πρόγραμμα τελείως, το NER 300 γι' αυτό σας, εδώ σας δείχνω τις βασικές δυσκολίες ανάπτυξης ενός προγράμματος CCS, δέσμευσης και αποθήκευσης. Όταν μιλάμε για ανανεώσιμα έργα, ανανεώσιμης ενέργειας, έχουν, ε, παράγουν ενέργεια, εν συνεχεία πωλείται και τα έσοδα θα πρέπει να ε, δικαιολογούν μια, ένα επιχειρηματικό σχέδιο Έχουμε όμως και χρηματοδοτικά αλλά και λειτουργικά προσκόμματα, διότι για να ανακτήσουμε από τη στιγμή που αρχίζει η ανάκτηση μέχρι την αποθήκευση είναι πολύ πιο ακριβή η όλη διαδικασία από την ενίσχυση ETS. Αυτό είναι το μεγάλο πρόσκομα, το μεγάλο εμπόδιο. Είναι λοιπόν το μπαλάκι πηγαίνει στα χέρια σας να αποφασίσετε αν αξίζει ή όχι. Το, το, το άλλο θέμα που σας είπα είναι ότι χρειάζεται και συνέργεια με την υποδομή των μεταφορών. Μέχρι τώρα είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας σε προγράμματα point-to-point. -point. Τώρα τωρα όλα τα προγράμματα ενίσχυσης των προγραμμάτων αυτών χρηματοδοτούν συγγνώμη, ή μελετώνται από διάφορες γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν. άλλο ένα εμπόδιο. Λοιπόν, η μεταφορά δεν αποτελεί κεντρικό στοιχείο του όλου προγράμματος. Πώς λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε πυρήνες αποθήκευσης ή σταθμούς αποθήκευσης CCS χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης ε, των μεταφορών, της υποδομής μεταφορών. Θέλουμε επίσης βεβαίως να εμποδίσουμε τη διασυνοριακή μεταφορά και το dumping των αποβλήτων. Εφόσον λοιπόν θέλουμε λύσεις, αυτή τη στιγμή θα αναγκαστούμε να κάνουμε υπερσυνοριακή, υπερσυνοριακή αποθήκευση. Αυτό λοιπόν πρέπει να λυθεί το θέμα. Ε, τα προγράμματα CCS θα πρέπει να καλυφθούν, να εμπεδοθούν στο, στο πλαίσιο ETS ε, υπάρχει βεβαίως το πρόβλημα των διαρροών και το πρόβλημα των εκπομπών αργότερα, ας πούμε μετά από 20 χρόνια λειτουργίας μιας εγκατάστασης και μετά από άλλα 20 χρόνια θα κλείσει η εγκατάσταση. Δηλαδή, μπορείς να πουλήσεις το διοξίδιο 5 ε, ευρώ τον τόνο, αλλά να έχεις ε, την, τον κίνδυνο, εάν υπά, διαφυγεί η εκπομπή, θα πρέπει να διαρροεί και η έκκληση, συγγνώμη, θα πρέπει να πληρώσει 50 ευρώ τον τόνο αργότερα, με τις ζημίες δηλαδή. Ε, και θα καταλήξω λέγοντας ότι η από την πλευρά της βιομηχανίας πρέπει εμείς να λάβουμε υπόψη το όλο κόστος και τα ε, εμπόδια στην μεταφορά και στην αποθήκευση. Αυτοί που λειτουργούν την πλευρά του EMP ε, δεν σκέφτονται αυτά τα προβλήματα, αλλά η ζημιά που μπορεί ενδεχομένω να επέλθει από τι διαρροέ και την έκκληση του διοξιδίου του είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε τώρα μία ακόμα παρουσίαση όσον αφορά το βίο αέριο δεύτερης γενιάς από την κυρία Άζα Μπούρμαν. Έχετε το λόγο. Σα eh, Σας ευχαριστώ. Προερχόμαι από το Gothenburg της ε, Σουηδίας και ασχολούμαι με ένα project το οποίο ονομάζεται Gobi Gas. Βλέπετε εδώ πέρα την βασική μονάδα επεξεργασίας ε, του ε, σχεδίου αυτού στο Gothenburg. Στο πάνω μέρος της εικόνας βλέπετε ότι όντως ασχολούμεθα με τον ανανεώσιμο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την χρήση άνθρακα. Μέσω λοιπόν του σχεδίου αυτού Θέλουμε να καταδείξουμε ότι μπορεί να παράγει κανείς βιοαέριο χρησιμοποιώντας διάφορα προϊόντα, εντελώς διαφορετικά προϊόντα τα οποία μπορούν να πάρουν τη μορφή ενέργειας. Πρόκειται λοιπόν για ένα σχέδιο σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορα στάδια. Έχουμε εξεργαστεί το σχέδιο αυτό με το Πανεπιστήμιο του Γκότεμπορκ, καθώς επίσης και με το Open University. Η μονάδα μας στο Gothenburg είναι πολύ μεγάλη και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο στάδιο του σχεδίου αυτού. Καταφέρνουμε να παράγουμε βιοαέριο της τάξης των 20 ΜΒ και στο δεύτερο στάδιο βλέπετε τη μονάδα εκείνη η οποία θα επεξεργαστεί το σχέδιο εκείνο το οποίο επελέγει στα πλαίσια του NER 300. Στόχος μας είναι η συνεχής βιώσιμη παραγωγή βιοαερίου Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι εταίροι που έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι ανάλογο στα πλαίσια του προγράμματος NER 300. Εμείς προσπαθούμε να παράγουμε βιοαέριο όχι σε μικρή κλίμακα όπως οι υπόλοιποι εταίροι, αλλά σε βιομηχανική κλίμακα, σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Στη συνέχεια το βιοαέριο αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί στους βασικούς κόμβους του ενεργειακού δικτύου προκειμένου να φτάσει στη συνέχεια στους μεμονωμένους καταναλωτές. Υπάρχουν πάντως πολλοί καταναλωτές και πάρα πολλοί παράγοντες στην αγορά που ενδιαφέρονται για την παροχή αυτή βιοαερίου και για τις ενεργειακές εφαρμογές του. Πέρα από το βιοαέριο ασχολούμεθα και με τα βιοκαύσιμα αλλά και αυτά θέλουμε να τα παράγουμε στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο. Βλέπετε λοιπόν ότι θα έχουμε ένα φόρτο παραγωγής της τάξης των 8.000 ωρών. Θέλουμε ουσιαστικά να παράγουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τόσο μεγάλη κλίμακα που θα μας επιτρέπουν και να τις χρησιμοποιούμε στα πλαίσια του επίσημου ενεργειακού δικτύου, αλλά και να καταφέρουμε να αντλήσουμε επικοδομητικά διδάγματα από το όλο εγχείρημα. Η μονάδα αυτή που βλέπετε στη Σουηδία είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας και θα αυξήσει την παραγωγή μας κατά 10%. Στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος βλέπετε ότι πενταπλασιάζεται η παραγωγή μας και χρησιμοποιούμε εξελιγμένη τεχνολογία τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο στάδιο. Στόχος μας είναι η ε, βιομηχανική εμπορική εφαρμογή της ενέργειας αυτής. Βλέπετε εδώ πέρα πάλι μια μονάδα παραγωγής ε, στο Gothenburg. Στα αριστερά το πράσινο βέλος δείχνει τη μονάδα παραγωγής ε, του πρώτου σταδίου του προγράμματος, ενώ με το δεύτερο βέλος βλέπετε την δεύτερη μονάδα παραγωγής, όπου, ε, στην οποία θα εφαρμόσουμε ουσιαστικά το δεύτερο στάδιο του προγράμματος. Ξεκινήσαμε στα τέλη του 2011 το πρόγραμμα συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 2012 και πλέον έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί πλήρως. Βλέπετε εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες από την ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής και μετατροπής ενέργειας. Βλέπετε εδώ πέρα διάφορους χώρους αποθήκευσης της ενέργειας. Βλέπετε το, την υποδομή αεροποίησης. Εδώ πέρα βλέπει μια φωτογραφία πριν από τρει εβδομάδες όταν αρχίσαμε τις εργασίες μας, όταν αρχίσαμε να λειτουργούμε επίσημα ουσιαστικά. Το γεγονός αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και ελπίζουμε τα πράγματα θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχικές μα εκτιμήσει. Βλέπετε εδώ πάλι μια φωτογραφία. Δεν προχωρούμε εδώ πέρα σε καύση αερίου. Βλέπετε όμως ότι όντως παράγεται από τη μονάδα αυτή παραγωγής αέριο, αέριο. Βλέπετε επίσης τις διάφορες μονάδες συμπίεσης και τον τρόπο που στη συνέχεια μεταφέρεται στο επίσημο δίκτυο διανομής ενέργειας. Είχαμε μια πολύ σημαντική υποστήριξη από την Ενεργειακή Αρχή της Σουηδίας μετά από την σχετική έγκριση που μας δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε χάρη στην χρηματοδότηση που μας δόθηκε μέσα σε 1,5 χρόνο να καταλήξουμε σε κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα. Όπως σας είπα, τα πρώτα αποτελέσματα είναι θετικά. Θεωρούμε ότι το σχέδιο αυτό είναι απόλυτα καινοτόμο και σε καμία περίπτωση δεν στρεβλώνουμε τον ανταγωνισμό με τη δική μας συνεργασία. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο στάδιο του project Gobigas. Πάλι εδώ έγινε ένα έλεγχο μια ανάλυση του δεύτερου σταδίου του προγράμματος αυτού. Η έκβαση της ανάλυσης αυτής ήταν πάρα πολύ θετική. Μπορούμε πέρα από την εμπορική εφαρμογή του σχεδίου αυτού να προχωρήσουμε και σε μία υλοποίησή του πάλι σε βιομηχανική μεγάλη κλίμακα. Ξέρετε ότι δυστυχώς βρισκόμαστε πάντα αντιμέτωποι με τις πολύ χαμηλές τιμές των ορυκτών καυσίμων, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει το δικό μας το έργο, την πρόωθηση των δικών μας προϊόντων, αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και επίσης υπήρξε και μια κάποια καθυστέρηση στην επίτευξη των αρχικών στόχων που είχαμε θέσει. Θεωρούμε ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει μια ξεχωριστή αγορά για το βιοαέριο. Βλέπουμε όμως ότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αντιμετωπίζουμε ένα πολύ έντονο ανταγωνισμό. Ξέρετε ότι στη Σουηδία επιδοτείται το φυσικό αέριο. Επιδοτούνται επίσης πολλές ε, συμβατικές μορφές ενέργειας, καθώς επίσης και τα ορυκτά καύσιμα, πράγμα το οποίο μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Εμείς πάντως είμαστε αισιόδοξοι και θεωρούμε ότι πολύ γρήγορα θα αρχίσει να λειτουργεί πλήρως η μονάδα αυτή παραγωγή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε για αυτήν σας την ε, παρουσίαση και την την εμπειρία αυτή που είναι τόσο πρόσφατη και τόσο σημαντική την οποία μας ε, περιγράψατε. Τώρα, ο κύριος ε, Μπερνάρ Ντελπές για την αποθήκευση ενέργειας. Σας δίνω αμέσως το λόγο. Euh, bonjour, <coughs> messieurs. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θα σας παρουσιάσω αυτά που μπορούμε να πούμε σήμερα από την άποψη της αποθήκευσης ενέργειας. Εγώ εκπροσωπώ έναν οργανισμό που ονομάζεται ΕΑΖΕ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ένωση για την Αποθήκευση Ενέργειας, όπου υπάρχουν διάφορα μέλη, κυρίως εταιρείες, από το βιομηχανικό κλάθο και ερευνητικά κέντρα και αυτή η Ένωση έχει την ιδιαιτερότητα να εκπροσωπεί όλους τους φορείς που ασχολούνται με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Την ΕΝΤΕΕΦ, την ΕΡΟΝ, την RWE, η Έλια επίσης συμμετέχει καθώς και κατασκευαστές πολλών υλικών. Η ΕΟΝ, η Alstom και ούτω καθεξής. Είμαστε μια μεγάλη ένωση λοιπόν για την αποθήκευση ενέργειας που στόχο έχει να δώσει μια συνέπεια και συνοχή στις διαφορετικές θέσεις που υπάρχουν. Για την αποθήκευση είναι απλή η αρχή, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας όταν δεν είναι πολύ ακριβή και χρήση της όταν έχει ε, ανέβει τιμή πολύ σύντομα. Λοιπόν, αυτή είναι και η χρησιμότητα της αποθήκευσης. Για την ηλεκτρική ενέργεια, να πω ότι σπανίως αποθηκεύεται με ένα μόνο μέσο, αλλά πάντοτε υπάρχει χρήση κάποιου μεταβατικού ε, μέσου για την αποθήκευση, το ευρωπαϊκό τοπίο προς την αποθήκευση. Έχει να κάνει χαρακτηρίζεται από κάποιες βασικές πρωταρχικές τάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την πολύ σημαντική ανάπτυξη των ε, περιστασιακών ε, βέβαια ε, αλλά υπαρχουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η βιομάζα. Το είπαμε και προηγουμένως. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παράγεται αν υπάρχει αιωλική ενέργεια, άνεμος ή ήλιος. Είναι λοιπόν περιστασιακή η παραγωγή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για πολλές χώρες της Ευρώπης και η παρουσία τους ε, έχει μεγάλες ε, συνέπειες και στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Από τεχνικής τώρα πλευράς. Βλέπετε τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Στο διάγραμμα φαίνεται η ζήτηση που έχει να κάνει με, τις, ε, με την με το σύνολο της θερμικής παραγωγής. Δηλαδή, τι γίνεται όταν η αιωλική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν φτάνουν. Έχουμε υπολογίσει όλο αυτό το ποσοστό με βάση το κλιματικό έτος, άνεμος, ήλιος και βροχοπτώσεις. Μέσα σε μία ημέρα βλέπουμε ότι αν διαιρέσουμε την ημερήσια κατανάλωση δια τις 24 ώρες έχουμε 30 γιγαβάτ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίπεδο ένωσης δηλαδή. Με, 150, από 30, με, διακύμαση από 30 έως 150 γιγαβάτ αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας αναλόγως. Τώρα, στις ανανεώσιμες βλέπουμε ότι περνάμε από 10 έως 30 γιγαβάτ ε, βιωσιμότητας μέσα σε μία ημέρα. Ανάλογα με τη θερμοκρασία και την ύπαρξη όχι ανέμου μέσα σε μία ημέρα μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη διακύμανση. Εάν πάρουμε τις υψηλότερες τιμές ε, ανανεώσιμων αιωλικής και ιαλικής, περνάμε στα 200 γιγαβάτ. Σας αφήνω εσείς να καταλάβετε πόσο ε, μεγάλα θέματα μπορεί να γύρει αυτή η μεγάλη διακύμανση. Το σύστημα λοιπόν, το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί ευελιξία. Αυτή την ευελιξία δεν μπορεί να μας την παράσχει μόνο η αποθήκευση, αλλά και τα λεγόμενα backup. Οι βοηθητικές λύσεις, ή το πώς θα διαχειριστούμε τη ζήτηση, η καλύτερη διασύνδεση των δικτύων. Αιωλική ενέργεια από τη Βόρεια Ευρώπη, λόγου ευρωπη λογω χαρη σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία. Ή το τι μπορούμε να πούμε σήμερα για την αποθήκευση. Ε, η σημασία της αποθηκευσής και το τι ευελιξία μπορεί να μας ε, παράσχει είναι ότι όλη αυτή η μοχλή μαζί στο μέλλον, όλα αυτά τα συστήματα στο μέλλον θα πρέπει να μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρικό δίκτυο ασφαλές και όχι ιδιαίτερα ακριβό. Η αποθήκευση λοιπόν. Η Ένωση μας ε, ασχολείται με όλες τις τεχνολογικές λύσεις για την αποθήκευση. Θα αναφέρω πολύ σύντομα αυτή που ονομάζουμε χημική ε, αποθηκευσή όπως το υδρογόνο με την εκτρόληση με ολική ενέργεια αποθηκεύω λοιπόν ε, η ηλεκτρική που είναι πολύ σπανιότερη η μηχανική, η πλέον γνωστή με υδραυλική ενέργεια 90% ε, της αποθηκευσής σήμερα στον κόσμο το νερό δηλαδή, το οποίο κατεβαίνει και μετά ανεβαίνοντας παρέχει πάλι ενέργεια, η θερμική ενέργεια και άλλες λύσεις. η θερμική επιτρέπει την παραγωγή θερμότητας όταν δεν είναι πολύ ακριβό το κόστος. Τώρα, από την πλευρά της Γαλλίας, Ξέρουμε ότι με την ε, ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να θερμαίνεται το νερό τη νύχτα όταν δεν είναι τόσο ακριβή ηλεκτρική ενέργεια και το πρωί να χρησιμοποιείται για τον ντους λόγω χάρη. Επίσης υπάρχουν ηλεκτροχημικές λύσεις, οι μπαταρίες δηλαδή που σήμερα έχουν αρκετά μεγάλη ανάπτυξη, ιδίως διότι υπάρχουν και τα ηλεκτροκινητά οχήματα. Υπάρχουν όλες αυτές οι τεχνικές λύσεις με δύο βασικούς τομείς εφαρμογής. Τις τεχνολογίες που παράσχουν ισχύ και αυτές που παράσχουν ε, ενέργεια. Ως προς την ε, ισχύ. Μιλάμε για όλες αυτές τις τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν ε, το να συνδυαστεί σωστά και να ξεροποιηθεί η ζήτηση με την αίτηση. Δηλαδή, να καλυφθούν σύντομες ανάγκες, ε, βραχυπρόθεσμες ανάγκες, άμεσα ή, ξέρω, ή λόγου χάρη η αποθήκευση ενέργεια τη νύχτα για να χρησιμοποιηθεί την ημέρα που είναι πιο ακριβή. Ως προς την, ε, έχουμε λόγου χάρη την, τις μπαταρίες, ενώ ε, με την ενέργεια, ενώ με την υδροελεκτρική, τη θερμική και τις υπόλοιπες λύσεις. Το διάγραμμα αυτό δεν θα σας πω στις λεπτομέρειες, απλώς δείχνει ότι η αποθήκευση είναι χρήσιμη σε όλα τα στάδια που ονομάζουμε ηλεκτρικού φόρτου για την παραγωγή, τη μεταφορά, την διανομή και τις υπηρεσίες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη βιωσιμότητα και πολύ μεγάλη χρησιμότητα από τις δυνατότητες της αποθήκευσης. Για τις ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσαμε εδώ να δώσουμε κάποια έμφαση. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε την ευελιξία της αποκεντρωμένης παραγωγής θα πρέπει να επιτρέψουμε στις περιστασιακές πηγές να μας δώσουν την απαραίτητη ισχύ. Επίσης θα πρέπει να περιορίσουμε τις αναταράξεις. Και οι ανανεώσιμες πηγές να περιορίζονται όταν υπάρχει πλεόνασμα και να αποθηκεύονται ε, απέναντι. Γιατί τώρα είμαστε σήμερα εδώ μπροστά σας και μιλάμε για την αποθήκευση γιατί είναι αυτό σημαντικό. Η αποθήκευση χρειάζεται τη στήριξη της ανάπτυξης και έρευνας και καινοτομίας. Γιατί, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλές αναδυόμενες τεχνολογικές λύσεις. Τεχνολογικές λύσεις που γίνονται ανταγωνιστικότερες από ότι είναι ελακτικές λύσεις. Ένα παράδειγμα, σήμερα οι μπαταρίες γίνονται ανταγωνιστικότερες για τη ρύθμιση των ε, συχνοτήτων στα ηλεκτρικά δίκτυα. Οπότε σε κάποια μέρη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη χρησιμοποιούνται οι μπαταρίες, χρησιμοποιούνται οι μπαταρίες για να υπάρξει η βασική ρύθμιση που χρειάζεται από τα ε, που χρειάζονται τα ηλεκτρικά εργοστάσια. Η έρευνα θα πρέπει μέσα σε μια διετία να ενισχυθεί περαιτέρω και θα πρέπει μέσα σε αυτή τη διετία να υπάρξουν και φορείς πρόθεσης για να είμαστε βέβαιοι ότι όλο αυτό το σύστημα θα μπορέσει να λειτουργήσει και στο μέλλον. Ξέρετε την περίπτωση του NER 300, αλλά είπαμε ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει και σε επίπεδο ρύθμιση στην Ευρώπη, γιατί από το διάγραμμα αυτό βλέπετε τι μεγάλες διαφορές υπάρχουν στις τιμές από την βασική ρύθμιση, εξισορρόπηση στην Ευρώπη, κάτι που δεν ευνοεί την ανάπτυξη της αποθήκευσης. Κατά τα άλλα, για τα μετέπειτα χρόνια, σύστασή μας είναι η αποθήκευση να γίνει μέρος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να αρχίσουν να αναπτύσσονται Μεγάλε χειρά παραδείγματα που χρησιμοποιούν την θερμική ιδίω αποθήκευση, την υπόγεια θερμική αποθήκευση, ώστε να υπάρχει μεταφορά εφόσον χρειάζεται καλοκαίρι ή χειμώνα. Να φτάσω στα συμπεράσματά μου. Μπορώ να σα πω ότι η αποθήκευση είναι ένα μέσο που ε, ουσιαστικά προσφέρει υπηρεσία σε όλη την αλυσίδα παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, ότι πρόκειται για νέα μέσα όπω οι μπαταρίε λόγω χάρη και ότι υπάρχει τέτοιο βαθμό χρησιμότητα που ε, ουσιαστικά θα μας επιτρέψει μεγάλες εξοικονομήσεις όπως το κόστος σε σχέση με τις σημερινές μεθόδους όπως χρησιμοποιούνται. Μπορούμε να αποφύγουμε την αύξηση λοιπόν του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας ε, να τρέχουμε στην αποθήκευση. Για κάποιους είναι μια τελείως νέα δραστηριότητα, αλλά έχει βιομηχανικό μέλλον στην Ευρώπη ο τομέας αυτός. Νομίζω ότι το NER300 που αφορά κυρίω τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην αποθήκευση, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα μέσο το οποίο είναι απολύτω αναγκαίο για να μπορέσουν οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια να συμπεριληφθούν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Παραγωγή Ηλεκτρισμού. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Ντελπέ. Ακούσαμε λοιπόν τρει ε, διαφορετικέ πραγματικότητε στην παρουσίαση τριών διαφορετικών πραγματικότητων και για τις ιδιαιτερότητες που έχουν και για τις προκλήσεις που παρουσιάζουν και θα δώσουμε τώρα το λόγο στο συνάδελ, στους συναδέλφους, στους εισηγητές και βεβαίως και τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, εμπειρογνωμονές μας γιατί ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι εμπειρίες που μας παρουσίασαν ε, κατά πρώτον μία παρατήρηση. Υπάρχει μια τεχνική δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα εξαιρετικά χρήσιμη. Η μετατροπή της βιομάζας σε, από την ε, σε φυτικά ε, παράγωγα το οποίο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο και για τα νερά αλλά και για την ε, γονιμότητα των εδαφών. Είναι ένα παράδειγμα του CCS που είναι ουσιαστικά στην πλευρά της ε, ενεργούς αντίδρασης και όχι της παθητικής. Μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των εδαφών. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο από την παρουσίαση της κυρίας Μπέρμαν είναι το εξής. Η τεχνολογική λύση που μας παρουσιάσατε είναι σημαντικότατη. Η ερωτήση μου λοιπόν είναι η εξή. Ουσιαστικά δημιουργείται πίσω από την ε, συμπίκνωση και εγώ έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να κατασκευαστούν περισσότερα εργοστάσια, μικρότερα εργοστάσια, για να καλύψουμε και το κόστος της μεταφοράς της ε, βιομάζας στα εργοστάσια. Εδώ για την αποθήκευση ενέργειας. Εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους αποσυμπυκνωτές υψηλής ε, ε, ισχύω, υψηλής τάσης, για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και με χρόνους ε, επαναφόρτισης που να είναι αρκετά σύντομοι. Έπειτα υπάρχουν και συστήματα αποθήκευσης ε, θερμότητας που και αυτά μπορούν να παρουσιάσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν χρησιμοποιηθούν σε εργοστάσια μικτής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, θέρμανσης διότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για την ε, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή να επιτρέπουν την αποθήκευση θερμότητας όταν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη από θερμότητα στη Γερμανία. Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα συνδυαστικού δικτύου, πολύ ενδιαφέρον και καλό θα ήταν να το κοιτάξουμε για να το χρησιμοποιήσουμε και αλλού. Πρόεδρος, πριν συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους, να παρακαλέσω να είμαστε κάπως σύντομοι γιατί είμαστε λίγο... Ε, έχουμε καθυστερήσει λίγο και Επίσης να πω στους ε, ομιλητές μας εδώ, στο Προεδρείο, ότι κάποιοι συνάδελφοι μου επισημαίνουν ότι θα θέλαν τις γραπτές ε, σημειώσεις από τις ε, ομιλίες σας διότι τους δώσατε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα παρακαλέσω λοιπόν και τη γραμματεία να μας φωτοτυπήσει τις ομιλίες για να τις δουν και οι συνάδελφοι. Ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ρώτησα και προηγουμένως γιατί χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια από την πρώτη στιγμή που αποφασίστηκε το NER 300 και την ανάθεση των έργων, των, των πρώτων αναθέσεων. Τέσσερα χρόνια χρειάστηκαν για να ε, συνδυάσουν όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς οι ε, κομισιόν. Όσον αφορά το πράσινο υδρογόνο, η πιο καινοτομική, ε, το πιο καινοτομικό στοιχείο είναι αυτό. Τώρα, εάν Εάν το NER λάβει προσφορές για προγράμματα NER 300, ε, λένε ότι ίσως δεν ήταν κατάλληλα όλα τα στοιχεία, όλες οι πτυχές ε, των προγραμμάτων αυτών. Ε, και η Κομισιόν εφόσον ε, είναι μυστικοπαθής όσον αφορά τις υποβολές αυτές των προτάσεων και ποιοι είναι υποβάλλοντες κλπ. κλπ. Δεν, τα πράγματα δεν προχωράνε. Χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία, περισσότερη διαφάνεια. Είπαμε ότι στο, μετά τον πρώτο γύρο υποβολής προτάσεων του NER300 παρουσιάστηκε ένα, μία αίτηση, μία πρόταση. Ε, είναι λοιπόν σωστή αυτή η αξιολόγηση της κατάστασης, καταλαβαίνουν τους περιορισμούς ε, μέσα στους οποίους έπρεπε να ενεργήσει η Κομισιόν, κανόνες είναι κανόνες. Αλλά θέλω να ρωτήσω, εάν είχε εγκριθεί και είχε πάρει όλες τις κατάλληλες άδειες το πρόγραμμα πράσινου υδρογόνου, δεν θα είχαμε δει καλύτερα αποτελέσματα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μαρίτα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Όσον αφορά την εγκατάσταση, τη μονάδα στο Γκότεμπεργκ. Ε, από ό,τι κατάλαβα, είπατε ότι η εγκατάσταση αυτή, η μονάδα αυτή είναι έτοιμη, αλλά είναι πειραματικό, πειραματική μονάδα. Πώς μπορεί τώρα να μετατραπεί σε μία ε, λειτουργική κανονική μονάδα και μάλιστα μεγαλύτερης κλίμακας έτσι ώστε να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και τι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν μέσα στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να έχουμε μία πρόοδο μεγάλης κλίμακας και τέτοιες μονάδες μεγάλες στο μέλλον. Ε, μήπως είναι το, πρόβλημά σας ότι ε, ε, η εξάρτησή σας από την ενέργεια προέρχεται κυρίως από δάση. Ε, ε και παραδείγματο χάρη εμείς έχουμε δυσκολίες όσον αφορά την ενεργειακή παραγωγή από τα δάση της Βραζιλίας και της Ινδονησίας όπου υπάρχουν τεράστια προβλήματα Υπάρχει λοιπόν διαφοροποίηση στη χρήση των δασών για ηλεκτρική ενέργεια στη Σουηδία έναντι της Βραζιλίας και της Ινδονησίας. Ποια είναι η κατάσταση σε εσάς. Ο κύριος Κέλλη. Thank you very uh, Κύριος Κέλλη, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλους τους συζητητές για τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους. Θα ήθελα πράγματι να τις είχαμε γραπτός για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όλα τα επίκαιρα θέματα που ε, μας αφορούν για τους κανονισμούς και το πλαίσιο γενικά. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές, με ενδιαφέρον ιδιαίτερα, διότι πιστεύω ότι αρχίζει μια αλλαγή της, ε, του κοινού, μια αλλαγή προσέγγισης και νοοτροπίας των πολιτών εγώ νομίζω ότι πολύ περισσότεροι έχουν αντιρρήσεις τώρα από ό,τι θα είχαν πριν από μερικά χρόνια και υπάρχουν και μεγάλες αντιρρήσεις όσον αφορά την οπτική επίδραση των ανεμογεννητριών και των ελικών πάρκων που πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι αντιρρήσεις. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα του κόστους που είναι των παραδοσιακών πηγών ενέργειας το ασυνεχές, το στοιχείο του ασυνεχούς. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, εάν αναπτύξουμε τον τομέα της αποθήκευσης και για να, να έχουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερου περιθωρίου χρήσης το πρωί ας πούμε, θα είναι πιο ελκυστικές, θα γίνουν πιο ελκυστικές οι εναλλακτικέ πηγές και πιο οικονομικά βιώσιμες. Η πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ. Είμαι πολύ ευτυχής που άκουσα όλες αυτές τις εισηγήσεις και τα επιτεύγματα που μπορέσατε να μου παρουσιάσετε έτσι ώστε καταλαβαίνουμε ότι ανανεώσιμες πηγές είναι ένα στοιχείο του μέλλοντος. Ένας ομιλητής είπε ότι η αποθήκευση είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα και η μεγαλύτερη πρόκληση, ιδίως σε ώρες εχμής ζήτησης της ενέργειας. Εγώ νομίζω πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο CCS, δέσμευση δηλαδή και αποθήκευση, και να αποδείξουμε ότι αυτή η μέθοδος είναι καλή για το μέλλον. Και μπορεί παρόλο που τώρα δεν χρησιμοποιείται ο άνθρακας όσο παλιότερα, ίσως θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο στο μέλλον όταν αναπτυχθεί το, το όλο project δέσμευσης και αποθήκευσης. Επίσης, όσον αφορά τις εναλλακτικέ πηγές, έχουμε διευρύνει τα τεχνολογικά συστήματα, παραδείγματο, χάρη αιωλικά ανεμογεννήτριες, αιωλικά πάρκα κλπ. Και, παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα και άλλες μέθοδοι για την αποσύσκευση της ενέργειας και τα σημείωσα από τις παρουσιάσεις σας. Γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε τις εισηγήσεις σας εγγράφως να μας τις ε, διανύμετε, διότι έτσι θα μπορέσουμε να, δείξουμε πώς το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 και το NER 300 μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Ο κύριος Καντσάν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τις παρουσιάσεις σας. Θα αναφερθώ στην παραγωγή κυρίως. Μολονότι βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε και να διατηρούμε, να αποθηκεύουμε την ενέργεια και να τη χρησιμοποιούμε όταν είναι αναγκαία. Αυτό το είπαμε και πριν από λίγο, ιδίως στα πλαίσια της παρουσίασης για την αποθήκευση που ακούσαμε. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω κάποιες σχετικές ερωτήσεις. Σήμερα όταν σπαταλούμε ενέργεια, όταν πετάμε τελικά ενέργεια χωρίς να την έχουμε αξιοποιήσει, ακριβώς επειδή δεν τη χρειαζόμαστε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ως προς αυτό, ποιες είναι οι δικές σας συμβουλές, έτσι ώστε να καταφέρνουμε κατά περίπτωση και σύμφωνα με συγκεκριμένα αιτήματα και ανάγκες ενέργειας να χρησιμοποιούμε την ενέργεια. Όχι απαραίτητα το ποσό της ενέργειας που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη μέρα ή τη νύχτα, αλλά να είμαστε σε θέση να δώσουμε ενέργεια όταν αυτή ακριβώς απαιτείται, όταν αυτή είναι αναγκαία. Και από τις μεθόδους παρουσιάσατε ποια προσφέρει περισσότερα εχέγγυα, περισσότερες διασφαλίσεις και κατά την άποψή σας ποιος είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε τις νέες αυτές δυνατότητες από πρακτικής πλευράς διότι έχω την εντύπωση ότι επιμένουμε πάρα πολύ στο ζήτημα της παραγωγής ενώ πέρα από τις μεθόδους που παρέχουν τα περισσότερα χέγγια, καταφέρνουμε τελικά να παράγουμε σημαντική ποσότητα ενέργειας, η οποία στη συνέχεια όμως δεν χρησιμοποιείται, δεν αξιοποιείται. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας και θα ήθελα να ακούσω και την απάντησή σας. Ο κύριος Γκέμπελς έχει το λόγο. Euh, Κύριε Πρόεδρε, σας το συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι μου δώσετε το, το λόγο, δεν κατάλαβα ότι είπατε το όνομά μου. Κυρία Πρόεδρε, με έχετε καλύψει. Όντως θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις, καθώς και η παρουσίαση του κυρίου Ντελπές. Μας δόθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες Πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα, με συγχωρείτε, όσον αφορά τη διακύμανση της ενέργειας, την συνεχή αυτή παροχή ενέργειας. Και τα στοιχεία αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά την παροχή όλων αυτών των διαφορετικών μορφών ενέργειας. Ακούσαμε και κάποιες εκτιμήσεις, κάποιες μελλοντικές προβλέψεις και τα δεδομένα αυτά νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να καταφέρουμε να συζητήσουμε επικοδομητικά μελλοντικά όλες αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, Λίκη Πρόεδρος. Κορέρα κάπου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους μας για τις παρουσιάσεις τους καταφέραμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μάθουμε πολύ χρήσιμα πράγματα. Ωστόσο εκπλήσωμαι όταν βλέπω ότι στο ζήτημα της αποθήκευσης της ενέργειας δεν υπάρχει κανένα άμεσο πρόγραμμα το οποίο να πορεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο να εστιάζεται επακριβώς την αποθήκευση ενέργειας. Η αποθήκευση ενέργειας εντάσσεται απλώς ως επιμέρους πρόγραμμα σε γενικότερες κατηγορίες προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με το πρασίνισμα της οικονομίας ε, ή με την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν χαίρει της προσοχής που θα έπρεπε να έχει, όπως μας είπε ένας παρουσιαστής. Ακούσαμε στην τελευταία παρουσίαση ότι υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις στην παροχή ενέργειας, ότι πολλές φορές η διανομή της ενέργειας είναι ασυνεχής. Ξέρετε ότι ε, αν συνεχίσουν αυτές οι αναταράξεις στην παροχή ενέργειας και αν τελικά συνεχίζουμε να έχουμε πολύ σημαντική παραγωγή φυσικού αερίου στο μέλλον, δεν αρκεί απλώς να επικεντρωνόμαστε σε κάποια σχέδια και σε κάποια projects όπως στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με συγκεκριμένα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την αποθήκευση ενέργειας και όχι μόνο με τα προγράμματα αυτά τα οποία έχουν κάποιον θετικό οικονομικό αντίκτυπο. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν για ποιο λόγο έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο πρέπει η αποθήκευση να αποτελεί απλώ επιμέρου τμήμα ενό γενικότερου ευρωπαϊκού προγράμματο και για ποιο λόγο δεν αποτελεί ξεχωριστό πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο το λόγο. Προέρχομαι από μια περιφέρεια της Ευρώπης που έχει την υψηλό ποσόστοση, την υψηλότερη ποσόστοση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Και έχουμε πάρα πολλές εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και έχουμε μία, ένα υπερβολικό πλεόνασμα παροχής ενέργειας και έχουμε αποθηκευτικές, ε, ε, έχουμε δυνατότητες μετατροπής της ανανεώσιμων, των ανανεώσιμων πηγών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φυσικό αέριο. Το ερώτημά μου είναι στην ενεργειακή πολιτική, στην πολιτική αποθήκευση, έχουμε συνδέσει δύο στοιχεία. Μείωση του διοξιδίου του άνθρακος το έχουμε συνδέσει με την απέτηση της βιομηχανίας για ανανεώσιμες πηγές. Αυτά τα δύο στοιχεία τα έχουμε συνδέσει. Στη δική μου περιφέρεια λοιπόν αυτό σε τι οδήγησε. Οδήγησε στην υψηλότερη ποσόστοση ε, χρήσης ανανόσιμων πηγών, αλλά ταυτό, ταυτόχρονα και αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα. Η δέσμευση και αποθήκευση, το CCS, το οποίο βεβαίως ε, ε, εξαρτάται πάρα πολύ από την ανοχή και έγκριση του κόσμου, ε, αναρωτιέμαι πώς θα δεχθεί οι πολίτες μας, πώς θα δεχθούν τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Καλό αυτό από τη μία πλευρά για την ενεργειακή επάρκεια, την από την άλλη πλευρά όμως διαβλέπουμε και υψηλούς κινδύνους. Ε, ε, διαφοροποιείται τους κινδύνους ανάλογα με τις εγκαταστάσεις. Και δεύτερον, είσαστε σε θέση από επιστημονικής πλευράς να συγκρίνετε και να αξιολογήσετε τις ε, διαφορετικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή ξεκινάτε από την προσέγγιση ότι πρέπει οπωσδήποτε ε, να ξεκινήσουμε με τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης και να μην μελετήσουμε τις άλλες ε, πτυχές. Αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, ας ακούσουμε τώρα τις απαντήσεις από τους καλεσμένους μας. Δίνω καταρχάς το λόγο στον κύριο Ντελγκάτο Ρώσα. Έχετε τρία λεπτά ο καθένας και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους ομιλητές. Λοιπόν, στα τρία αυτά λεπτά θα επικεντρωθώ στο σημαντικότατο αυτό ζήτημα της ευελιξίας στα πλαίσια του προγράμματος NER300 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και γενικότερα. Το πράσινο υδρογόνο όντω αποτέλεσε θύμα της έλλειψης ευελιξίας στα πλαίσια του προγράμματος NER300. Κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να πάρει μία απόφαση αναφερόταν σε συγκεκριμένα άρθρα του κανονισμού με αποτέλεσμα τελικά να έχουμε διάφορα λειτουργικά προβλήματα και προσκόμματα, τα οποία θα είχαν στη συνέχεια πρόβλημα στην ε, ίδια τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, Επενδύσεων διαμεσολαβούσε για την χρηματοδότηση και κάθε φορά αναφερόταν στον κανονισμό του ΝΕΡ 300. Δεν είμαι λοιπόν απόλυτα σίγουρος αν θα μας βοηθούσε περισσότερη ευελιξία για, τον, για το πράσινο υδρογόνο. Πάντως υπήρχαν σίγουρα διάφορα προβλήματα χρηματοδότησης. Για ποιο λόγο τώρα έχουμε αυτή την έλλειψη ευελιξίας στα πλαίσια του ΝΕΡ 300. Διαχειριζόμαστε τους πόρους των κρατών μελών με τρόπο ανταγωνιστικό. Δεν είναι εύκολο λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, να έχουμε απόλυτη ευελιξία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάζει όποτε θέλει τους κανόνες και να προσαρμόζεται στις επιμέρους περιστάσεις. Θα έλεγα βέβαια ότι θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από την εμπειρία αυτή, τουλάχιστον για τα μελλοντικά προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτήσουμε. Να δούμε για αυτά μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιδείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία και να δώσουμε μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Όπως σας είπα όμως υπάρχει και το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος. Τουλάχιστον στην δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων προσπαθούμε να δούμε ακριβώς ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει ο κάθε εταίρος στις προτάσεις που υποβάλλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδα επίσης ότι υπήρχαν και κάποιες παρερμηνίες θεωρώ ότι όλοι έχουμε αντλήσει και από αυτές διδάγματα, είτε πρόκειται για τα κράτη-μέλη, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τους φορείς αυτούς καθ' αυτούς. Πάντως ε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση στο ζήτημα της ευελιξίας αν ε, συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε το πρόγραμμα ner R300 με πόρους των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ για την καλή χρήση του χρόνου. Ας ε, ακούσουμε και τους υπόλοιπους ομιλητές με τη σειρά που μίλησαν. Το, λόγο έχει ο κύριος Ζάκα Κιβίτε. Σας ευχαριστώ. Σας είπα ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε τις αποφάσεις της Ολλανδικής κυβέρνησης. Απαντώ λοιπόν έτσι τον κύριο Ντέιβις. Χρειάστηκε να συμμορφωθούμε με τις αποφάσεις της κυβέρνησης αυτής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε τελικά το πρόγραμμα το οποίο υποβάλαμε και το οποίο δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση. Σαφώς λοιπόν υπήρχαν κάποιες παρανοήσεις και δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουμε περισσότερες πληροφορίες που ενδεχομένως θα επέτρεπα στο σχέδιο αυτό να προχωρήσει περισσότερο. Αν υπήρχε μεταξύ μόνο μια πολύ καλή συνεννόηση, θα είχε εγκριθεί το πρόγραμμα αυτό και θα είχε δώσει ήδη κάποια αποτελέσματα. Τώρα όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό, νομίζω ότι χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα δέσμευσης και αποθήκευσης, το οποίο παράλληλα προσπαθεί να επαναχρησιμοποιήσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να δημιουργήσει συνέργειες. Πραγματικά κρίμα που δεν χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα αυτό και ελπίζω να πάτησα στην ερώτησή σας. Grazie. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπέρμαν. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις πρώτα τα όλα του κυρίου Πρόντι για το μέγεθος των εγκαταστάσεων. Στην Σουηδία και τη Φινλανδία έχουμε αρκετά τέτοια εργοστάσια. Με μεγάλη εκτογραμμή στις χώρες αυτές έχουμε πολλές ε, πολύ μεγάλη ποσότητα και διαθεσιμότητα φυσικών πρώτων υλών σε μικρή απόσταση. Μπορούμε λοιπόν πολύ εύκολα να μεταφέρουμε είτε συντηροδρομικός είτε δια της θαλασσίας οδού τις πρώτες αυτές ύλες. Αυτός προς την πρώτη ερώτηση. Μετά τέθηκε η ερώτηση για το τι γίνεται με το Γκέτεμπορκ και το μεγάλο εργοστάσιο εκεί. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και αυτό ένα υποδειγματικό εργοστάσιο, αλλά Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι εάν μας βοηθούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαμε και την ευκολία να περιορίσουμε την, ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να υπάρξει έτσι εναρμόνιση στις πτυχές της διαχείρισης. δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διάφορε χώρε έχουν και διαφορετικά επίπεδα χρηματοδότησης ή στήριξη, οπότε αυτό επηρεάζει και τον ανταγωνισμό. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από τότε που ελήφθη αυτή η απόφαση πριν από ένα χρόνο. Όταν έπεφταν οι τιμέ ε, των ορειτών ε, καυσίμων και ήταν τελείως διαφορετικά τα δικαιώματα εκπομπών και οι τιμέ τους. Ήταν διαφορετική η υπολογισμή μας ως προς τη χρηματοδότηση. Νομίζω πολλά προγράμματα λοιπόν και από το 1 er ER300 υποφελήθηκαν από αυτή την παράταση. Τώρα για το τι δεξιότητες θα, χρειαζόντουσαν, ε, θα χρειαζόταν η διαχείριση των ε, δασικών ε, καταλήπων η δασοκομεία στη Σουηδία είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία της χώρας και ήδη σήμερα χρησιμοποιούμε τα δασικά κατάλοιπα με τρόπο όσο το δυνατόν πιο βιώσιμο. Υπάρχουν όμως διαφορετικές ε, περιστάσεις και συνθήκες στις διάφορες χώρες. Εμείς θα παράγουμε κυρίως βιοαέρια, τα οποία ελπίζουμε να αξιοποιήσουμε στον τομέα των μεταφορών. Όμως σήμερα Χρειάζεται να υπάρξουν και κάποιες διασφαλίσεις για το, ε, από, για το τόπο προέλευσης των, ε, των πρώτων υλών, ώστε να υπάρξει και ε, ασφάλεια για το κοινό. Τώρα για την εξαέρωση γενικώς σε διαφορετικές χώρες υπάρχουν και διαφορετικέ πηγές. Είναι άλλε στην Αυστρία και άλλε λόγω χάρη σε εμά όπου μπορούμε να αντλήσουμε από τα πράσινα, από τις άλγες. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι από τον υπόλοιπο κόσμο έχουμε αυτή τη στιγμή ε, συνεργασία ούτε στη Σουηδία ούτε στη Φιλανδία Πρόεδρο, ευχαριστούμε και τελευταίο ο κύριο Ντελπέ διότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η δική του ομιλία. Μάλιστα. Για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας είδατε ότι υπάρχουν πολλαπλές λύσεις και θα πρέπει ο καθένας να προσαρμόζεται. Στην παρουσίαση που έκανα έδωσα έμφαση στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι σημαντική και η αποθήκευση ισχύω, όπως έλεγα όμως, γιατί οι ανανεώσιμες πηγές έχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια ε, εξισορρόπηση της ισχύω για να μπορεί να αξιοποιηθεί. Η αποθήκευση σε μπαταρίες ή σε, άλλα, ε, σε άλλες συσκευές όπως τα flywheel είναι πολύ σημαντικά. Πάντως, το αν αύριο θα μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε την ενέργεια που παράγεται, αυτό θα το απαντούσω ως εξή. Υπάρχουν δύο εναλλακτικέ οδοί. Υπάρχει το υδρογόνο, κάτι που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερως ε, στην Γερμανία λόγω χάρη, αλλά υπάρχει και η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λύση της ε, υδραυλικής άντλησης. Υπάρχει από πολλά χρόνια αυτό, όπως στη Γαλλία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, αλλά παράγει και θερμότητα σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή θερμαίνεται το νερό όταν υπάρχει λόγω χάρη πολλής άνεμος, αλλά θερμαίνεται όταν χρειάζεται να παραχθεί και ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε, ουσιαστικά, είναι αυτό που έλεγα εξ αρχή ότι πρέπει να προσαρμόζεται η παραγωγή στη ζήτηση. Νομίζω ότι η αποθήκευση είναι ο καταλληλότερο τρόπο να το πετύχουμε αυτό και η αποθήκευση θερμότητας είναι από τις πλέον υποσχόμενες λύσεις σε αυτό το τομέα. Και με το νερό, με τη χρήνη αξιοποίηση του νερού, αλλά και με άλλου τρόπου. Πολλέ έρευνε γίνονται σχετικά και νομίζω ότι είναι από τις ωραιότερε ε, τις προσφορότερες μάλλον λύσεις. Τώρα για την αποθήκευση τη νύχτα είναι σημαντικό με τα σημερινά δεδομένα. Όμως αν αναπτυχθεί και άλλο η ηλιακή ενέργεια, το κόστος μπορεί να μειωθεί. Οπότε θα υπάρχει μια ε, δευτερεύουσα ζήτηση η οποία μπορεί να είναι λιγότερο σημαντική από την ζήτηση της νύχτας. Η αποθηκευσή μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο τοπίο που θα διαμορφωθεί από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία όπως ξέρουμε διαφέρει από την ημέρα στη νύχτα, παραδοσιακά τουλάχιστον. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κάποιες φορές καθυστερώ να σας ε, πάρω το μικρόφωνο, διότι η ταλική μετάφραση καθυστερεί πάντοτε λίγο παραπάνω. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια, είμαστε μπροστά από, την, ε, από το πρόγραμμα, οπότε να δώσω στον κύριο δεν Ντερόζα τον λόγο για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα τη αποθήκευση. Ευχαριστώ, θα το αξιοποιήσω αυτό το εξτρά λεπτό που μου δίνετε, γιατί έγιναν πολύ σημαντικά σχόλια. Οι προκλήσει για την ενέργεια είναι πολλαπλέ. Δεν χρειαζόμαστε μόνο μία χρυσή συνταγή για ένα θέμα, αλλά χρειάζεται να συνδυάσουμε πολλά ενεργειακή αποδοτικότητα, αποθήκευση, ευφύη δίκτυα, εσωτερική αγορά. Αλλά η αποθήκευση πραγματικά είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Γίνονται πολλές έρευνες για την αποθήκευση, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το 2020, το Horizon 2020 θα μας επιτρέψει να δώσουμε μία θεώρηση για το μέλλον, αλλά μπορούμε με την αποθήκευση να καλύψουμε το κενό μεταξύ πιλωτικών προγραμμάτων και της τελικής απόδειξης. Ελπίζουμε πως ναι, αλλά η προβολή στο μέλλον θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να μελετήσουμε πολύ καλά την αποθήκευση. Η αποθήκευση ίσως δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα ως προς την πρόσληψη του κοινού όπως έλεγα. Δηλαδή δεν θα αρέσουν σε όλους ε, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον αλλοιώνουν το, ε, το, τοπίο. Συγγνώμη. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν μια χρυσή συνταγή, δεν είναι αυτή η αποθήκευση, αλλά σίγουρα αξίζει να την κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμεί. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτήν την ακρόαση, η οποία ήταν μέρο του προγράμματο εργασιών τη Επιτροπή μα. Την είχαν ε, ορίσει οι συντονιστέ. Νομίζω η ακρόαση αυτή ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για όλου. Ευχαριστώ λοιπόν του εισηγητέ μα, οι οποίοι μα παρουσίασαν τι χειροπιαστέ, συγκεκριμένε εμπειρίε του και στάθηκαν σε όλα τα σημεία με μεγάλη σαφήνεια και με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως το NER 300 και τα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικά παρόλο που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και αυτή τη στιγμή το οικονομικό μας σύστημα μετατοπίζεται προς ένα σύστημα ε, ενεργειακά συμβατικό με όλα αυτά. Πάντως πρέπει να δούμε και τις πτυχές της επένδυσης. Το θέμα της επένδυσης, των επενδύσεων λοιπόν, για να δούμε τι επενδύσεις χρειάζονται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επενδύσεις που ίσως να είναι ε, σοβαρές, αλλά με τον καιρό να μπορέσουν να δώσουν και τα ε, ωφέλη που ε, περιμένουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τις παρουσιάσεις σας. Η συζήτηση συνεχίζεται και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που μας παρακολούθησε σε όλη αυτή την ακρόαση. Ευχαριστώ. Il Μάλιστα, συνεχίσουμε λοιπόν. Εξετάζοντας τις κοινέ επιχειρήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Για την σχετική αυτή συζήτηση έχουμε στη διάθεσή μας μια μισή ώρα. Έχουμε τρεις ε, παρεμβάσεις ε, για τις πέντε διαφορετικές κοινέ επιχειρήσεις. Σήμερα το πρωί και το απόγευμα θα μιλήσουμε για το ΣΕΖΑΡ, καθώς επίσης και για τις ε, τέσσερις εταιρικές σχέσεις δημοσίου τομέα. Έχουμε εδώ και τους πέντε συναδέρφους εισηγητές, στους οποίους δίνω πέντε λεπτά στον καθένα για να μας παρουσιάσουν την έκθεσή τους. Ξεκινάμε με την συνάδελφο Ριέρα Μαντουρέλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι όταν οι κυβερνήσεις κόβουν τα κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη και επενδύσεις, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τα μέσα που ενθαρρύνουν ε, περισσότερες ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Και ακριβώς ε, αυτά τα κοινά προγράμματα μπορούν να βελτιώσουν τις επενδύσεις δεδομένου ότι προσφέρουν ένα πολυετές σταθερό πλαίσιο και έτσι μπορεί και ο βιομηχανικός τομέας, ο τομέας δηλαδή, να δεσμευτεί έναντι περισσότερων υποχρεώσεων. Θα Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να επιβάλλουμε μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ ε, των ε, κοινών προγραμμάτων δημόσιο-ιδιωτικό τομέα και να γίνουν περισσότερες δημοσιεύσεις υποβολής προτάσεων και να ε, διαδοθεί πολύ περισσότερο η ανάγκη και η ενίσχυση της έρευνας στην επιστημονική κοινότητα. Γι' αυτό έχουμε υποβάλει ένα μεγάλο αριθμό τρόπολογιών, όμως δεν έχω πολύ χρόνο και θα ήθελα να εστιάσω σε δύο συγκεκριμένα θέματα, σε δύο πτυχές που ε, πιστεύουμε ότι είναι πιο σημαντικές. Καταρχάς όσον αφορά ε, την πρωτοβουλία καινοτομικών ε, ε, φαρμακών και τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτά έχουν άμεση σχέση με, την, τον προϋπολογισμό. Έχω μιλήσει με τους συζητητές και των άλλων κοινών προγραμμάτων και θα εφαρμόσουμε το 12,5% ε, το οποίο ε, μας υποχρέωσε το Συμβούλιο να εφαρμόσουμε στο πρόγραμμα ΠΚΑΦ2 διότι πιστεύουμε ε, μέσα στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ε, το Συμβούλιο μας έχει περιορίσει σε αυτό τη μείωση κατά 12,5% και θέλουμε να εφαρμόσουμε διακρατικές πρωτοβουλίες να ε, συνεργαστούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε δίκτυο και γι' αυτό δεν θέλουμε ε, τα προγράμματα αυτά να ε, έχουν ε, αρνητική επίπτωση, να υποστούν ζημία λόγω των περικοπών του Συμβουλίου. Ε, θέλουμε τα προγράμματα αυτά, το pkf 1 και το pkf 2 να χρηματοδοτηθούν επαρκώς. Ε, με βάση τα κριτήρια αριστείας. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η, να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης πολλαπλασιαστικότητας ε, και πολλαπλασιασμού των προγραμμάτων αυτών. Θα θέλουμε ένα νέο δείκτη έντασης, έρευνας ε, και τεχνολογίες. Αυτός ο δείκτης έχει εισαχθεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ε, όσον αφορά τώρα την ε, πολιτική για ε, τα φάρμακα αυτά, έχουμε την έκθεση OD και το Κοινοβούλιο ζητάει τη χρηματοδότηση ε, των προγραμμάτων υπό το προγραμμα pkf ΠΚΑΠΑΦ2 να χρηματοδοτούνται υπό μία δέσμη κριτηρίων. Αυτό συνάδει και με τη γενική πολιτική των κοινών προγραμμάτων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Ε, τα, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι έχουν ακόμα ε, μεγάλες αμφιβολίες όσον αφορά την εφαρμοστέα πολιτική στα πλαίσια των ΣΔΙΤ και όλα τα μέλη του IMI θα ήθελαν να ε, υιοθετηθεί μία προσέγγιση χωρίς εμπόδια, χωρίς προσκόμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι έχω υποβάλει τροπολογίες για την παγίωση ε, της Επιστημονικής Επιτροπής ως το κύριο σώμα, αρμόδιο σώμα, για να εξασφαλίσουμε ότι όλες ε, οι φορείς, οι φορείς θα λάβουν τα απαραίτητα ε, κονδύλια τα οποία χρειάζονται σε αυτή την πάρα πολύ ευαίσθητη, στον ευαίσθητο τομέα. Ευχαριστούμε την κυρία Μαντουρέλ. Τώρα ο κύριος Φανίστερόη. Προέρχομαι, μόλις μπήκα στην αίθουσα, θέλετε να πω κάτι συγκεκριμένο για την, ε, τα προϊόντα της ε, βιοιατρικής ε, και τα προανταγωνιστική βιοτρική. Τι θέλετε να κάνω ή μόνο, μόνο αυτά τα οποία βασίζονται στη βιοτική. Εντάξει, αυτό όπως είναι στην ημερήσια διάταξη δηλαδή. Λοιπόν, αυτή τα, η προανταγωνιστική βιοτική και τα προϊόντα είναι το καινούριο μας παιχνιδάκι, το καινούριο μας ε, μωρό και τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πλαίσιο και ε, βλέπω, διαπιστώνουμε ότι και στον αρμόδιο οικονομικό τομέα υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός, μεγάλη προθεμία σύμπραξης. Εάν ξεκινήσουμε εξ αρχής μόνο με ένα δισεκατομμύριο, τότε θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε ένα προαπλησιαστή ε, στην οικονομική πλευρά, στην βιομηχανική πλευρά και θα καταλήξουμε σε 2,8 δισεκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το έναυσμα πολλαπλασιάζεται εν συνεχεία λόγω της προθυμίας του τομέα. Αυτό είναι πάρα πολύ, ένα πολύ θετικό στοιχείο και πιστεύω ότι μπορούμε να ενεργήσουμε γρήγορα, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια καλή προετοιμασία και μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, στον τομέα αυτόν. Έχω λίγες ε, τροπολογίες ε, να παρουσιάσω. Το μόνο που πιστεύω είναι ότι πρέπει να μάθουμε από την εμπειρία των άλλων. Χρειαζόμαστε μία ενσωματωμένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και τις προόδους της έρευνας και ανάπτυξης της, ε, του τομέα και έχουμε μεγάλες πιθανότητες επιτυχίες. Να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο αυτό τον κύκλο. Εάν γίνουν περικοπές στις προκλήσεις της κοινωνίας, society challenges, τότε πιστεύω ότι αυτές οι περικοπές πρέπει να γίνουν αναλογικά και όχι να είναι μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλους τομείς. Πρέπει να υπάρχει ε, ίση κατανομή των περικοπών και κάθε ε, πρόγραμμα, ε, για, κάθε πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα μπορούν να έχουν τη δική τους ανάπτυξη. Ε, λυπάμαι αν μειωθούν τα κονδύλια από το πλαίσιο, αλλά τουλάχιστον να είναι οριζόντιες οι περικοπές. Οι αναλογίες πρέπει να είναι ίδιες, σωστές και δίκαιες, διότι εμείς στοχεύουμε στο να λάβουμε 2,8 δισεκατομμύρια. Ε, έχω περιοριστεί πολύ στις τροπολογίες, αναφέρομαι σε ορισμένες στις εξαιρέσεις ακόμα και στην απαλλαγή νομίζω πρέπει να υπάρχουν ακόμα ο, ο, εκρεμή ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί με τις άλλες πρωτοβουλίες αλλά όπως σας είπα θα ακολουθήσω μια πολύ περιορισμένη και μετριοπαθή στάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βανιστερόη. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Σέλερ. Πέντε λεπτά. Κυρίες και κύριοι, το ορίζοντας 2020, ε, το πρόγραμμα ορίζοντας 2020 έχει ε, διαμορφωθεί και τώρα ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες. Η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 2 συνολικά θα καλύπτει 9 δισεκατομμύρια, ένα σημαντικό στοιχείο. Όμως είναι περίεργο που αυτό το κονδύλι ε, λαμβάνει τόσο διαφορετικά ονόματα, τόσο διαφορετικούς ορισμούς. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία πακέτο με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Το λέω αυτό επειδή βασιζόμενοι στις συνθήκες έχουμε μια διαφορετική κατάσταση με τα διάφορα προγράμματα ΣΔΙΤ, ε, δηλαδή σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια συμφωνία πακέτο. Το επιχείρημά μας πρέπει να είναι ότι ο χρόνος πιέζει, ε, βρισκόμαστε στη φάση διαβούλευσης ε, και αν χρειαστούν ε, εξουσιοδότηση πράξη τότε θα πρέπει σαφώς να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα θέματα στην, ε, ως πακέτο για να μπορέσουμε να δεχθούμε τις παρεκκλήσεις και την έκδοση κατεξαίρεση πράξεων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του χειρισμού σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο θα είναι ότι θα μπορέσουμε να δούμε αποτέλεσμα ε, και να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα πριν λήξει η θητεία του Κοινοβουλίου. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, η πρωτοβουλία, το PKF είναι πολύ σημαντικό για τις ε, νέες ε, για και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στη δημόσια υγεία, μείωση εκπομπών κλπ. Πιστεύω ότι το PKF2 είναι, θα επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα και όπως το προηγούμενο, το ε, Clean Skies, θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Εγώ στην έκθεσή μου αναφέρουμε όχι σε συγκεκριμένες θέσεις, αλλά ε, στην ε, περιθώριο καινοτομίας και βελτιώσεων που υπάρχουν. Η Κομισιόν στο Clean Sky 2 σημειώνει ότι οι βελτιώσεις είναι πολύ σημαντικές και σε ορισμένε περιπτώσεις οι βελτιώσεις ήταν 60%, ε, ε, δεύτερον, η Κομισιόν πιστεύει ότι μπορούμε να παίξουμε ένα μεγαλύτερο δραστήριο ρόλο στο Clean Sky 2 και να επιτύχουμε μεγαλύτερες συνέργειες Επίσης, ε, όσον αφορά το Clean Sky 2, υπάρχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερο περιθώριο διαπραγμάτευσης από πλευράς Κοινοβουλίου. Υπάρχουν ακόμα μερικά θέματα που πρέπει να τα συμφωνήσουμε. Καταρχάς, ε, ο προϋπολογισμός. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και εδώ να βρούμε μια λύση πακέτο και πιστεύω ότι η μείωση του προϋπολογισμού κατά 12,5% θα γίνει, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός γενικού συμβιβασμού όλων των προϋπολογισμών και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων όχι επειδή θέλουμε να ξεκινήσουμε μια πολιτική διαμάχη αλλά όπως σας είπα και πριν για να υπάρχει μια ισορροπία ιδίως όταν το μεταφράσετε σε προκλήσεις διότι πολλοί τομεί είναι υπέρ της του προϋπολογισμού για το Clean Sky 2 αλλά και για ε, την έρευνα σε άλλους ε, τομείς όπως τις μεταφορές. Εάν λοιπόν δούμε τα ε, παράλληλα προγράμματα όπως το ΣΕΖΑΡ μαζί με το Clean Sky 2 και άλλα προγράμματα μεταφορών και έρευνας ε, πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να περιληφθούν σε ένα πακέτο. Επίσης την περιέλαβα το στοιχείο της μεσοπρόθεσμης αναθεωρη... αξιολόγησης, ενδιάμεσης αξιολόγησης η οποία δεν θα περιλαμβάνει μόνο την αξιολόγηση του προγράμματος ε, καθεαυτού, αλλά μία εις βάθος ε, αξιολόγηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών. Όσον αφορά τώρα την χρονική περίοδο θα θέλουμε να τη μειώσουμε ο, μέχρι το 2020 έτσι ώστε να ευθυγρομιστούμε με τον ορίζοντα 2020. η συνέργεια μεταξύ ε, ορίζοντας 2020 και Clean Sky 2 ε, θα οδηγήσει σε μία απλούστευση των διαδικασιών, διότι θα υπάρχει μία μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος 4 ετών, μεγαλύτερη από ό,τι υπήρχε στο Clean Sky 1. Θα έχουμε λοιπόν δύο παρόμοια προγράμματα αλλά με διαφορετικούς κανόνες χρηματοδοτικής συμμετοχής, ε, ε, διαφορετικό πλαίσιο, δηλαδή διαφορετικές κυβερνήσεις που συμμετέχουν κλπ. Και τέλος, αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι αυτή η μεταβατική περίοδος να διευρυνθεί ακόμα περαιτέρω για κάθε πρόγραμμα. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι εξετάζουμε μια πιο ε, παράλληλη προσέγγιση, μια πιο κοινή προσέγγιση με τα διαρθρωτικά ταμεία για τις επενδύσεις κυρίως. Δεν θα θέλαμε μείωση ε, και θα θέλαμε να ε, συνεχιστεί αυτή η θετική στάση της Κομισιόν και όσον αφορά τον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων. Ξέρω ότι αυτό επιβάλλει διοικητικό κόστος, αλλά δεν, δεν μπορώ να τα παραβλέψω όλα αυτά, γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια κονδύλια. Και για να καταλήξω θέλουμε ε, να υιοθετήσουμε ένα μια ευρύτερη προσέγγιση να προσθεθούν, δηλαδή να συμμετάσχουν περισσότερα κράτη-μέλη στο ορίζοντα 2020 όσον αφορά δηλαδή τη χρήση κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη από τα διαθροτικά ταμεία και δεύτερον από τη δική μας πλευρά ε, να υπάρχει μία ε, ρήτρα δικαιούχων, ε, εκείνων ναι, και για το Clean Sky 2 και όσον αφορά την αξιολόγηση και την απαλλαγή θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία ιδέα πώς θα γίνει αυτή η αξιολόγηση και ε, απαλλαγή. Ε, θα πρέπει να έχουμε μεμονωμένες απαλλαγές και όχι η απαλλαγή των προγραμμάτων να ενσωματωθεί στην ευρύτερη απαλλαγή του προϋπολογισμού και των διαδικασιών της Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε κύριε Έλερ. Ξέρετε ότι για την συζήτηση αυτή προβλέπονται ακόμα 30 λεπτά. Εξ αποστάσεως τώρα πρέπει να συγχαρούμε την συνάδελφό μας Κολάρσκα Μπομπίνσκα, η οποία όπως ξέρετε έγινε υπουργό για ζητήματα επιστημονικά στην Πολωνία. Συγχαρητήρια λοιπόν. Είμαι σίγουρη ότι θα τις διαβάσουμε κατά κάποιον τρόπο τα συγχαρητήρια μας αυτά. Και ο κύριος Ρούμπικ θα την αντικαταστήσει για την έκθεση που θα μας παρουσίαζε σήμερα. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό σημάδι αυτή η ανταλλαγή απόψεων που λειτουργεί θαυμάσια μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μας συνέβαλαν ε, πολύ θετικά ε, στην διαμόρφωση αυτού του πλαισίου για το μέλλον. Ε, και μάλιστα αυτό το πλαίσιο πρέπει να είναι σταθερό ε, ε, ιδίως για τη φετινή χρονιά και η μετάβαση από τα προηγούμενα προγράμματα πέρσι, η σταθερή μετάβαση σε ένα πλαίσιο φέτος ήταν πάρα πολύ σημαντική, δεδομένου ότι καταβάλαμε πάρα πολλές προσπάθειες να επιτύχουμε αυτό το σταθερό πλαίσιο και είδαμε τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται για τα, ε, για τα έργα δημοσίου, για τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα ΣΔΙΤ. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συνέργεια η οποία προβλέπεται στον ορίζοντα 2020 και να την ε, αναπτύξουμε περαιτέρω, ιδίως στους ε, διαφόρους τομείς, ε, όπως ας πούμε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει ορισμένες και να μελετήσει ορισμένες ενεργειακές καινοτομίες, επίσης τα θέματα της κατάρτισης ε, στην έρευνα και τεχνολογία, ε, το θέμα της επαγγελματικής ε, κατάρτισης και εξέλιξης, πληροφορική, όλοι αυτοί οι τομείς της τεχνολογίας και θα πρέπει να, να τύχουν της κατάλληλης ενίσχυσης στην εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να διδάσκονται ε, τα τελευταία δεδομένα για να μπορούν να ε, επωφεληθούν και από ε, εμπειρίες άλλων χωρών είναι καλό λοιπόν ότι έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας και ξέρουμε ότι η, ασφα... ηλεκτρονική ε, ασφάλεια διακυβέρνησης, το e-government και τα διάφορα ε, στοιχεία προστασίας ε, δεδομένων είναι πολύ σημαντικά γιατί δεν θα πρέπει να μειώνουν ή να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό έτσι ώστε Όλο το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα εκατομμύριο όπως ελέγχθη θα δοθεί από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, εκεί που για μένα υπάρχει κάποια επιφύληξη είναι γιατί τα διοικητικά, οι διοικητικές δαπάνες είναι τόσο διαφορετικές στα διάφορα προγράμματα έχουμε ας πούμε διοικητικό κόστος που υπολογίζεται σε 6% και σε άλλες πτυχές είναι ε, πάνω από 6% γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η διακύμανση του διοικητικού κόστους πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την αύξηση των διοικητικών δαπανών κατά 10% και αν υπάρχουν περιθώρια μείωσης. επίση, το Ευρωπαϊκό επιστημονικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να δώσει ορισμένες ενισχύσει, ορισμένα grants και αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν με το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο ε, έρευνα για να ε, ξεκινήσει μία νέα πρωτοβουλία από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης αξιολόγησης ε, προτάσεων και χρηματοδότησή τους. Όλα αυτά τα προγράμματα πρέπει να αξιολογηθούν με μεγάλη προσοχή διότι θα αντιμετωπίσουν την απαλλαγή και ορισμένα από τα προγράμματα αυτά είναι πολύ μεγάλα ε, και υπόκεινται στην άμεση, στον άμεσο έλεγχο του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται μία ανακοίνωση της Κομισιόν ε, και μία επικοινωνία, μία διαβούλευση για να δούμε πώς θα γίνει ο χειρισμός αυτού του τομέα για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Ίσως να χρειαστεί η εισαγωγή ενός, ε, μιας νέας διαδικασίας. Αλλά γενικά πιστεύω ότι αυτή η νέα διαμόρφωση των ΣΔΙΤ ε, θα είναι λίαν ωφέλιμη, λίαν πλεονεκτική για μας και θα ε, δώσει, ε, δραστηριοποιήσει αγορές οι οποίες για το μέλλον μας είναι πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρούμπικ. Η τελευταία παρέμβαση θα είναι από τον κύριο Τόντοροφ Παναγιόντοφ από τους φιλελεύθερους. Έχετε το λόγο κύριε Παναγιώτοφ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ σύντομα να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσής μου για ένα κανονισμό του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή επιχείρηση Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2. Υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία αναφέρω στο σχέδιο έκθεσης. Χαιρετίζω καθαρά, καταρχάς με συγχωρείτε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία της κοινή αυτής επιχείρησης για τα επόμενα δέκα χρόνια. Θεωρώ ότι μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να ασχοληθούμε με κάποιες πολύ σημαντικές πτυχές των κυψελών καυσίμου και του υδρογόνου. Η κοινή επιχείρηση Κυψέλε καυσίμου και υδρογόνου δείχνει το δυναμικό που έχει τόσο το υδρογόνο όσο και οι κυψέλε καυσίμου, ότι μπορούν να αποτελέσουν μετατροπή ενέργεια στην Ευρώπη για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια, να μειώσουν τι βλαβερές εκπομπές και να τονώσουν τη μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινή επιχείρησης που διεξήχθη το 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέδειξε ότι η κοινή αυτή επιχείρηση έχει με επιτυχία υπηρετήσει μέχρι σήμερα ως μια πλατφόρμα για τη δημιουργία στερεάς εταιρικής σχέσης προκειμένου να ενισχυθεί ο βιομηχανικός τομέας και ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών. Έτσι λοιπόν στην εκθεσή μου συνιστώ να χρησιμοποιήσουμε την επικοδομητική αυτή εμπειρία από το πρώτο πρόγραμμα και για την επόμενη δεκαετία. Το υδρογόνο είναι ένας φορέας ενέργειας, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα καθαρό καύσιμο και αποτελεί ουσιαστικά μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Έχει πολλές εφαρμογές και μπορεί να προσφέρει βασικές λύσεις στις πιο μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή ως τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την έξυπνη ανάπτυξη οι κυψέλες καυσίμου μπορούν με τη σειρά τους να δώσουν μια εναλλακτική μορφή ενέργειας στα ορυκτά καύσιμα, να εξασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια και να μειώσουν την εξάρτησή μας από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η χρησιμοποίηση τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τη διαθεσιμότητα κάποιων ε, βασικών πρώτων υλών, όπως ε, κάποια συγκεκριμένα σπάνια μέταλλα, όπως το λίθιο. Η έλλειψη των πρώτων αυτών υλών μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον πρόβλημα στη χρησιμοποίηση και την ανάπτυξη των κύψελών καυσίμου και του υδρογόνου και των σχετικών τεχνολογιών. Έτσι λοιπόν στόχος της δεύτερης κοινή επιχείρησης θα πρέπει να είναι η έρευνα και η ανάπτυξη καθώς επίσης και οι καινοτόμες στρατηγικές που να έχουν ως στόχο να βρεθούν εναλλακτικές πρώτες ύλες για την ανάπτυξη των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο η χρήση των δύο αυτών νέων μορφών ενέργειας θα βιώσιμη. Η εμπειρία από την πρώτη κοινή επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα θετική όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τις δημιουργίες θέσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης είχαμε κατά μέσο όρο μία 10% αύξηση στον ετήσιο κύκλο εργασιών, 8% μέση αύξηση στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, 6% ετήσια αύξηση στις θέσεις απασχόλησης και 10% ετήσια αύξηση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε εταιρείε του κλάδου αυτού. Συνιστώ επίσης στην έκθεσή μου να δοθεί μια απολογή, απαλλαγή με συγχωρείτε για τη διαδικασία αυτή όσον αφορά τη χρηματοδότηση και να συνεχιστεί η χρηματοδότηση όπως και στο παρελθόν. Η παράταση της κοινή αυτής επιχείρησης στέλνει ένα πολύ θετικό μήνυμα περαιτέρω δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω ανάπτυξη των κυψελών καυσίμου και του υδρογόνου. Θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε ένα σύστημα κυψελών καυσίμου και υδρογόνου πιο βιώσιμο και πιο ανταγωνιστικό και θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την ανάπτυξη και την παγκόσμια ανάπτυξη των νέων αυτών μορφών ενέργειας. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα έχουν πολύ θετικές επιπτώσεις, κοινωνικές, τεχνολογικές, πολιτικές, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε επιμέρους περιφέρειες και πόλεις. Θεωρώ λοιπόν ότι η κοινή αυτή επιχείρηση Κυψέλης, καυσίμου και υδρογόνου πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να συνεχίσει να εμβαθύνει περισσότερο σε ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης και θα πρέπει να βασιστεί ήδη στα πρώτα θετικά αποτελέσματα που έχουμε από την πρώτη κοινή επιχείρηση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να υποφεληθούμε από τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να δώσουν οι νέες αυτές μορφές ενέργειας για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο Οντί, ο οποίος αντικαθιστά την κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία λεπτά για κάθε παρέμβαση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, συγγνώμη από πλευρά τη κυρία Γκροστέτ, αλλά είχε βουλευτικέ υποχρεώσει στην χώρα τη. Να συγχαρώ την κυρία Ρία Μαδουρέλ για την αφοσίωσή της και το έργο της και δύο-τρεις προσωπικές παρατηρήσεις για το σύνολο του φακέλου. Πρόκειται για την πρωτοβουλία καινοτόμα φάρμακα με πολύ σημαντικό απολογισμό. Ε, στηρίζουμε την πρωτοβουλία του ΕΛΚ και αυτήν την κοινή επιχείρηση ιδιωτικού δημόσιου τομέα για την Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία με δύο δις ευρώ κύκλο Η περίοδος θα ε, παραταθεί ε, από το 2014 έως το 2020, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό στοιχείο. Όμως για την τροπολογία 11 της κυρίας Μαντουρέλ. Να πω, η πρόταση αύξησης ε, των κλινικών δοκιμών των κοινοτόμων φαρμάκων είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να παραμείνει ως έχει στη διατύπωσή του είναι κάπως ασαφή. Στη 12 προτείνεται για τις ε, παραγωνισμένες ασθένειες να υπάρξει καλύτερος εντοπισμός, όμως να μην απαριθμηθούν ακριβώς, ώστε να μην δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μια ή στην άλλη πάθηση νόσου. Για την τροπολογία 31 ζητάτε μεγαλύτερη συμμετοχή από την εισηγήτρια να φροντίσουμε το κριτήριο της αριστείας να είναι το πρωταρχικό. Στην τροπολογία 32 υπάρχουν οι προανταγωνιστικές, ε, οι πρόδρομες μάλλον δραστηριότητες που ζητούνται από την ε, εισηγήτρια εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε να επιδέχουμε πάντα το κοινοτόπο αποτέλεσμα. Στην ε, τροπολογία 21, 30 και 51 και 50, συγγνώμη, προτείνεται από την εισηγήτρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τι συστάσει τη ε, ομάδα εργασία για την υγεία μέσα στο πλαίσιο του προγράμματο ε, Horizon 2020. Όμω η ομάδα αυτή ακόμη δεν έχει συσταθεί. Διερωτώμεθα λοιπόν πω είναι κάπω περίπλοκο να υπάρχει μια τέτοια μνήμα. Τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική τη άποψη για την μείωση, την περικοπή στον προπολογισμό, εδώ είμαστε αρκετά διχασμένοι, διότι θεωρούμε ότι είναι ένα αρνητικό μήνυμα. Φανεί κάτι τέτοιο από την πρόταση. Τώρα για την μεταφορά από τον ε, προπολογισμό ναι, αλλά οι δείκτες των επιδόσεων να είναι ρεαλιστικοί και να ενισχυθούν οι παρακολουθήσεις και οι έλεγχοι. Από προσωπικής άποψης, εγώ υπήρξα εισηγητής για το, πρόγραμμα, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, την αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Είχαμε δει όλη τη βιοθητική και την ε, και βασική δομή και κοιτάξαμε κατά πόσον υπήρχαν οι απαραίτητες νομικές δομές σε κάθε κοινή επιχείρηση. Εδώ να σας πω ότι θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Υπάρχουν κοινέ επιχειρήσεις που είναι πρότυπα, υποδειγματικές διεθνώς για, τον, για τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Όμως έχουμε χάσει πολύ χρόνο για να μην χωρίς να έχουμε δει ε, ως βουλευτές τι κάνει το 80% αυτών των κοινών επιχειρήσεων και να μην μπορούμε να δώσουμε και απαντήσεις στους πολίτες. Ας προσέξουμε πολύ λοιπόν τι κάνουμε και κατά πόσο πολλαπλασιάζουμε αυτές τις προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει ως νομική βάση την ε, κανονισμό του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα δώσει μόνο τη σύμφωνη γνώμη του. Λυπάμαι, αλλά δεν το βρίσκω δίκαιο αυτό. Έχει δαπανηθεί πολύ χρήμα, έχουμε εργαστεί για τι συμβαστικέ λύσει πολύ σκληρά. Τη στιγμή λοιπόν τη σύμπραξη με τι επιχειρήσει μα παραγωνίζεται. Θα θέλαμε να καταλάβουμε τι εξήγηση δίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτι άλλο στο οποίο θα είμαστε αμετακίνητοι και να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι τη Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποσπάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ε, ε, απαλλαγή για τι κοινέ αυτέ επιχειρήσεις. Να θυμίσω ότι το ηλεκτικό συνέδριο και απευθύνουμε και στον Πολ που ήταν εισηγητή για την Επιτροπή Προπολογισμών. Εξέφρασε ενδιασμού για την οικονομική διαχείριση αυτών των κοινών επιχειρήσεων. Σε αυτή τη φάση το να μα ε, αποσπά αυτή την αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα καθήκον ελέγχου τη εκτελεστική εξουσία από την πλευρά του Κοινοβουλίου το βρίσκω παράδεκτο. Θα έπρεπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί επισήμω ότι θα λάβει υπόψη τι τροπολογίε μα, ιδίω για την απαλλαγή και του ελέγχου και μέσω του εκπροσώπου της. Διότι μας παίρνεται από τα χέρια μια αρμοδιότητα η οποία μας οφείλεται. Αναρωτιέμαι κατά πόσον έχετε το δικαίωμα να κάνετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Οντί, ο οποίος μίλησε και ως κύριος Οντί και εκ μέρους της κυρίας Γκροστέτ. Και τώρα η κυρία Άντρες Μπαρέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτές οι κοινέ επιχειρήσεις υπό το πρόγραμμα πλαίσιο έχουν ως στόχο να εδραιώσουν προγράμματα τεχνολογίας, να ενισχύσουν τα κοινά προγράμματα δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και είναι πάρα πολύ σημαντικές επιχειρήσεις. Θέλουμε να ενισχύσουμε την καινοτομία ε, στον βιομηχανικό τομέα και υπάρχει μεγάλος ο ενθουσιασμός. Η βιοιατρική είναι πάρα πολύ σημαντική ε, και χρειαζόμαστε ε, εδώ ε, ε, εγγυήσει ότι όλα τα, αυτά τα πράγματα είναι ανακυκλώσιμα, αυτά τα προϊόντα της βιοιατρικής είναι σωστά, είναι ασφαλή, είναι ανακυκλώσιμα και χρειάζεται να εξασφαλίσουμε μία ισορροπία όσον αφορά την αηφορία των οικοσυστημάτων όπως έχει τονιστεί σε πολλές άλλες εκθέσεις. Πράγματι, πολλές πρωτοβουλίες ε, ε, αναπτύσσονται, εξελίσσονται. Ο εισηγητής ε, αναφέρεται στο στοιχείο του ενθουσιασμού. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση σε όλες τις κοινέ αυτές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στο τομέα της βιο, βιομηχανικής, των προϊόντων της βιοιατρικής της βιοβιομηχανίας. Και συμφωνώ με τον κύριο Οντί. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε συμμετοχή και το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλέκεται, πρέπει να ε, συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Ε, θα υποβάλουμε βεβαίως ε, τροπολογίες εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και αυτός οι τροπολογίες εστιάζονται στην συνοχή με το πρόγραμμα πλαίσιο ορίζοντας 2020. Επίσης, οι τροπολογίε εστιάζονται περισσότερο στην περιφερειακή ανάπτυξη και στο περιφερειακό στοιχείο, στην αξιολόγηση και αναθεώρηση των προγραμμάτων και στο ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί τα προγράμματα. Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι σωστή, ε, δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον και Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εξετάζουμε και να εγκρίνουμε ή όχι τη χρήση δημοσίων κονδυλίων. Τη χρήση των κονδυλίων. Ευχαριστούμε την κυρία Μπαρεσανδρέα, ο κύριος Τζόνσον. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Είμαι σκιώδης εισηγητής... στο πλαίσιο ε, το, της προανταγωνιστικής βιοιατρικής και των προϊόντων της ε, και συμμερίζουμε αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής. Επίσης συμφωνώ με όλα τα προλεχθέντα σήμερα διότι είναι σημαντικό ε, να, να κινηθούμε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αλλά έχω ορισμένες απορίες, ορισμένα ερωτήματα μόλις ε, άκουσα αυτά τα οποία είπαν οι κύριοι Έιλερ και Βαν Μίσελρο και συμφωνώ μαζί τους. Αναφέρθηκαν στη δυνατότητα πολλαπλασιασμού, τον, ε, πολλα, τον πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ε, δηλαδή, ε, να υπάρχει ένα, μια αλφα συμμετοχή η οποία συνεχεία να πολλαπλασιαστεί. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συντονισμένη συμφωνία και με τα άλλα ε, ταμεία, παραδείγματος χάρη τα ταμεία της Ένωσης πρέπει να δούμε σε μια συντονισμένη διαβούλευση πού μπορούν να συμμετάσχουν τα κράτη, πού μπορούν ο δημόσιος δηλαδή τομέας και πού ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να μπορέσουμε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε και όσο το δυνατόν περισσότερο ε, αποτέλεσμα, απόδοση να έχει δική μας συμμετοχή. Μία άλλη συζήτηση που κάναμε στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μην ξεχνάμε αυτό το στοιχείο, πρέπει σοβαρά να ληφθεί υπόψη και η συμμετοχή τους. Διότι πολλές φορές η υπερβολική καινοτομία δημιουργεί εμπόδια, προσκόμματα σε μικρές επιχειρήσεις. Τρίτον, να μην ξεχνάμε τις προκλήσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Να εντοπίσουμε καινούριε ευκαιρίες, να τις εκμεταλλευτούμε, να χρησιμοποιήσουμε νέες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε συνεχώς να έχουμε κατά νου την αηφόρο ανάπτυξη. Είχα κάνει μία ε, πρόταση της καλύτερης, της βέλτιστης χρησιμοποίησης των προϊόντων της δασοκομείας. Εν κατακλείδη, έχω θετική προσέγγιση, συμφωνώ με αυτές τις προτάσεις των δύο εισηγητών και θα παρουσιάσω συγκεκριμένες τροπολογίες. Ευχαριστούμε, συνάδελφος Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω το ακόλουθο. Δεν θέλω να επαναλάβω τα λόγια των συναδέλφων. Απλώς θα πρέπει προφανώς να αντλήσουμε από την ε, πείρα που έχουμε ε, συγκεντρώσει από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και με στόχο το Horizon 2020. Θέλουμε να είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα αυτό και να μην ε, το καταβαραθρώσει το προβολικό διοικητικό άχθο. Ω εισηγητή για τα θέματα του υδρογόνου και της ε, Για το υδρογόνο λοιπόν, να πω ότι είδαμε το παράδειγμα του 7ου προγράμματος πλαισίου ότι ε, το διοικητικό άρθρο ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ε, οι επιχειρήσεις έτειναν να παραμένουν εκτός διότι καταλάβαιναν πόσο θα επιβαρυνθούν. Χρειάζεται όμω και έλεγχο για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Όπω είπε ο συνάδελφο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διάμεσε ε, αναθεωρήσεις και εκθέσει για να υπολογίζουμε την επιτυχία των διαφόρων προγραμμάτων και το πώ προχωρούν. Επίση, οι εταιρικέ σχέσει, οι κοινέ επιχειρήσει μάλλον δημοσιοδιοτικού τομέα, είναι μια πολύ σημαντική ε, εναλλακτική οδό για να προωθούνται οι ερευνητικέ δραστηριότητε. Ω ε, σκιώδη εισηγητή, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω και να διευκολύνω τη διάδοση των ε, συμπερασμάτων που μπορούμε να αντλήσουμε από το πρόγραμμα πλαίσιο, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν και θα κάνω ό,τι μπορώ για να συμβεί αυτό. Έχουμε παρόμοιες μέρημνες για το Horizon 2020 και θα πρέπει οποιοδήποτε προβλήματα παραμένουν να απελευθούν, ώστε η πορεία της έρευνας να είναι ανεμπόδιστη και να στοχεύει τις ερευνητικές δραστηριότητες και μόνον να επικεντρώνεται στην ουσία. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι πεπισμένο ότι το Horizon 2020 είναι ουσιώδου σημασία για την ανάπτυξη τη έρευνα στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο, ο συνάδελφο Μπραζίνα. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω και ο δισηγητή για τις εκθέσεις αυτές, συγκεκριμένα για το υδρογόνο και τις κυψέλευς καυσίμου, να πω ότι θα πρέπει να συνεχιστούν όσα ξεκίνησαν ε, με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, διότι ήταν πολλά υποσχόμενες τεχνολογικές λύσεις που είχαν βρεθεί εκεί. Δεν είναι μόνο το θέμα αν θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα την αποδοτικότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα άλλο, κάτι άλλο που είναι επίση σημαντικό είναι τα εφηδίκτια λόγου χάρη ή η χρήση της υδραυλικής ενέργειας, το αν θα υπάρξει καύση υδρογόνου ή το πώς θα λειτουργούν ακριβώς οι κυψέλευες καυσίμου. Είναι θέματα καθοριστικά για το μέλλον όλα αυτά να τονίσω απλώς μία πτυχή, μία από τις πολλές στις οποίες θα μπορούσα να σταθώ, ο κλάδος των ε, κυψελών καυσίμου και του υδρογόνου έχουν τεράστια σημασία από την πλευρά της διοργάνωσης των επιχειρήσεων. Για την ώρα δεν έχουμε ισχυρού όμως ε, πρωταγωνιστές στον επιχειρηματικό χώρο της Ευρώπης. Δείτε τι έγινε με το Clean Sky. Είχαμε ισχυρούς εταίρους οι οποίοι μπορούσαν και να χρηματοδοτήσουν σε μεγάλο βαθμό. Όμως για τις κυψέλες καυσίμου έχουμε μια δραστηριότητα που τώρα ξεκινά τα πρώτα της δηλάβηματα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί. Νομίζω το βασικότερο πρόβλημα θα είναι η συγχρηματοδότηση. Η συγχρηματοδότηση από την πλευρά του κλάδου των εταιριών, του μηχανικού κλάδου. Συμφωνώ λοιπόν με του συναδέλφου και είμαι στη διάθεσή του προκειμένου να συνεργαστούμε και να απαλείψουμε τι αρνητικέ πτυχέ που έχουν απομείνει από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και να δώσουμε μια όθηση στην πρωτοβουλία αυτή, η οποία είναι πολλά υποσχόμενη. Ευχαριστούμε ο συνάδελφος Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι έχουν εργαστεί σκληρά. Θα επικεντρωθώ στο Clean Sky για το οποίο είμαι σκιώδης εισηγητής της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Το Clean Sky 2 σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα που συζητούμε, έχει μια βιομηχανική ταυτότητα λίγο πιο συγκεκριμένη. Υπ' αυτήν την έννοια, αυτό που πιστεύω είναι ότι υπάρχει ανάγκη ο χρόνος που θα τρέχει αυτό το εγχείρημα να μην ε, περιοριστεί στον ορίζοντα του Horizon 2020 αλλά να του δοθεί ο ρυθμός που του χρειάζεται. Δηλαδή να διαφυλάξουμε τη βιομηχανική διάρθρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή χωρίς να ασκήσουμε χρονική πίεση. Επ' αυτήν την έννοια θεωρώ ότι είναι σημαντικό να φροντίσουμε την αλυσίδα ε, παροχής, supply chain, ε, το εργαλείο μέσω του οποίου θα μπορέσουμε να εμπλέξουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια με τρόπο εντονότερο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συχνά ε, μικρές ε, ούσες δεν συμμετέχουν ενεργά σε κάποιες πτυχές. Θα πρέπει λοιπόν ε, αυτό να είναι ένα βασικό στοιχείο της δράσης μας. Είναι και αυτές οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Η διαχείρισή μας λοιπόν σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης θα πρέπει να τους επιτρέψει και αυτές να ανθίσουν ε, στο χώρο αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο που θεωρώ σημαντικό είναι ότι μπορούμε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις κοινέ επιχειρήσεις, αυτές τις ε, κοινέ λοιπόν επιχειρήσεις, να τις διευκολύνουμε ε, εφόσον έχουν τα χαρακτηριστικά της διορατικότητας που θέλουμε και μπορούν να ενισχύσουν τη βιομηχανική διάρθρωση. Νομίζω ότι το στοιχείο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το θεωρήσουμε θεμελιώδες και αυτό της αλυσίδας παροχής όπως έλεγε. Αυτό θα είναι ένα από τα τεστ που θα δοκιμάσουν τα κατά πόσο μπορούμε να ενισχύσουμε τις δράσεις αυτές. Υπάρχει ανάγκη να δώσουμε στο ευρωπαϊκό βιομηχανικό κόσμο τα κίνητρα για να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, αλλά και σε ό,τι φορά την βιομηχανική διοργάνωση και διάρθρωση. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια επαναλαμβάνω την δέσμευσή μου, εποβάλλω τροπολογίες, προκειμένου να, μην να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του βιομηχανικού κόσμου αυτού καθεαυτού. Πρόεδρος, ευχαριστούμε συνάδελφος Καρβάλιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους ε, διάφορους εισηγητές για, τη, για τα σχέδια εκθεσή τους και την προθυμία τους να συνεργαστούν με όλους τους συναδέλφους. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύνολο των προτάσεών της και κάποια γενικά σχόλια για όλες τις κοινέ επιχειρήσεις. Κατά την άποψή μου, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα από τα σημαντικότερα θέματα θέματα που θα μας επιτρέψουν στην Ευρώπη να έχουμε ανάκαμψη και να ε, καθορίσουμε το μέλλον μας. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οι επενδύσεις των εταιριών στην έρευνα και ανάπτυξη είναι κρίσιμες για την ε, μελλοντική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εάν σταθούμε και δούμε το πρόσφατο τις πρόσφατες επιδόσεις των εταιριών ε, στην έρευνα και ανάπτυξη θα δούμε ότι το επίπεδο των επενδύσεων που διαρκώς μειώνεται από το 2008 κάπως ε, επανήλθε. Ε, από το 2004 για πρώτη φορά έχουμε και πάλι σε πρωταγωνιστικό ρόλο την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία στις δράσεις έρευνας και ανάπτυξης παγκοσμίως με την γερμανική Volkswagen. Προκειμένου λοιπόν να διατηρήσουμε τα επίπεδα καλού βιωτικού, τα επίπεδα μάλλον ε, κοινωνικής ευημερίας, θα πρέπει στις αυτοματοποιημένες βιομηχανίες, στην αεροναυπηγική, στη χημική βιομηχανία να διατηρήσουμε τον, τον πραγωταγωνιστικό μας ρόλο και να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος σε άλλους τομείς. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά και τα κλάστερς, καθώς και οι ε, εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή η αξιοποίηση των ε, άριστων ερευνητικών κέντρων και της επιστημονικής κοινότητας που διαθέτουμε είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον της οικονομίας της Ευρώπης. Επισημένω λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία στους συναδέλφους που ασχολούνται με τέτοια θέματα τα οποία είναι σημαντικότατα για την Ευρώπη. Είχαμε μία μείωση στη συμμετοχή των εταιριών ε, του μηχανικού κλάδου στο πρόγραμμα πλαίσιο. Τώρα έχει αυξηθεί η συμμετοχή τους. Οπότε, όπως προ, ως προ τον προπολογισμό χρειάζονται και τα απαραίτητα κονδύλια. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να υπάρξει εξισορρόπηση μεταξύ των κονδυλίων για τις κοινέ επιχειρήσεις και των υπολείπων. Όμως η βασική μου σύσταση είναι ότι θα πρέπει να απλουστεύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους κανόνες και να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ των ως τώρα ισχυόντων κανόνων και των ε, νέων που θα ισχύουν. Να μην υπάρχουν μεγάλες αλλαγές για τις εταιρείε μεταξύ των προηγούμενων και των ε, νέων κανόνων. Να υπάρχει μια σταθερότητα. Περισσότερη διαφάνεια επίση, περισσότερο ανοιχτό πνεύμα προ του νέου εισερχόμενου και το να ε, προωθήσουμε την αριστεία αλλά και να, να δώσουμε κίνητρα για τη συμμετοχή, καθώς και εξαγωγή σχέσεις ε, συνεργασίας με τα διευθυντικά ταμεία που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του Horizon 2020, αλλά και τα μεγαλύτερα βιομηχανικά σχέδια και εγχειρήματα που έχουμε να εξετάσουμε εδώ. Αυτά είναι τα σχόλιά μου για τις διάφορες τεχνολογικές κοινέ επιχειρήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τη συνάδελφο Καρβάλιο, η κυρία Φόρτ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ προηγουμένως γιατί έπρεπε να συμμετέχω σε τριμερείς διαλόγους για άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Βλέπω ότι όλοι εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά καθώς πλησιάζει το τέλος της κοινοβουλευτικής μας θητείας και σίγουρα τα ζητήματα που συζητάμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον της έρευνας και, για το της, της στην Ευρωπαϊκή Άνωση. Προσβλέπω λοιπόν να συνεργαστώ και με τους ηγητές και αυτής της Επιτροπής για τα ζητήματα αυτά, συνεργασία που έχω και με άλλους συναδέλφους σε άλλες επιτροπές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να προωθήσουμε γρήγορα, ιδίως τους φακέλους εκείνους για τους οποίους προβλέπεται συναπόφαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εγκρίνουμε όλες αυτές τις δέσμες, αλλά σε καμία περίπτωση να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στην όλη διαδικασία συναπόφασης και καθυστερήσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν γενικές περικοπές σε όλο τον προπολογισμό και ότι στη συνέχεια υπάρχει μια επιμέρους κατανομή στις κοινέ επιχειρήσεις. Δεν είμαι πεπισμένη ότι κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε λογικά. Άκουσα την κυρία Καρβάλιο που είπε ότι έχουμε πλέον και επιπλέον πόρους από τον ιδιωτικό φορέα. Σίγουρα αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε οριζόντιες περικοπές για αυτό το λόγο για όλες τις κοινέ επιχειρήσεις από τον κοινοδικό προπολογισμό, όπως άλλωστε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Θεωρώ ότι οι κοινέ αυτές επιχειρήσεις πραγματικά προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα την κοινή επιχείρηση Clean Sky. Θεωρώ ότι οι έλεγχοι και εξολογήσεις θα μπορούσαν να λάβουν χώρα προκειμένου τουλάχιστον από τεχνικής πλευράς να ξέρουμε ποιος αποφασίζει για την μεθοδολογία του ελέγχου, έτσι ώστε να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τα εμπιστευτικά δεδομένα των εταιριών που συμμετέχουν σε αυτή την κοινή επιχείρηση. Όσον αφορά τώρα την πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα, Ξέρετε ότι είχαμε και ένα πρώτο πρόγραμμα, μια πρώτη κοινή επιχείρηση, με την οποία πρέπει να συνάδει η δεύτερη αυτή κοινή επιχείρηση, το ένα πρόγραμμα να συμπληρώνει το άλλο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ποσοστώσεις όσον αφορά την εργασία που γίνεται σε τρίτε χώρε. Σε ορισμένε περιπτώσει ο στόχο μα είναι να καταφέρουμε να παράγουμε νέα καινοτόμα φάρμακα για συγκεκριμένες ασθένειες, παραμελημένες πολλές φορές ασθένειες, δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε συγκεκριμένε μόνο χώρε. Είναι σημαντικό να αποφεληθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τρίτε χώρε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνη και με τι χώρε αυτέ. Ορισμένοι λένε ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν θα πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένε κλινικέ δοκιμέ. Αν δείτε όμω κάποιε εξατομικευμένε ε, θεραπείες οι οποίες μπορεί να μην είναι πολύ ε, οικονομικά επωφελείς. Από την άλλη πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνονται γιατί ε, η ε, εξειδικευμένη κλινική δοκιμή στην τομέα, όπως για παράδειγμα στον τομέα των γονιδίων, μπορεί να βοηθήσει πιο διδεδομένες ασθένειες στην αντιμετώπιση τους, όπως για παράδειγμα την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Όσον αφορά το επιστημονικό τώρα πάνελ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σαφώς τις γνωμοδοτήσεις των επιστημών αυτών, χωρίς όμως να δημιουργήσουμε ένα ακόμα επίπεδο γραφειοκρατίας. Τώρα όσον αφορά την, τον προσιτό χαρακτήρα των φαρμάκων, πρέπει να εξασφαλίσουμε και πάλι ότι δεν θα δημιουργήσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια είναι πολύ σημαντική οποιαδήποτε θεραπεία προκύψει να μπορεί να είναι και προσιτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάντσιαν έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους συγητές. Θεωρώ ότι θα πρέπει πραγματικά να να αξιοποιήσουμε και να εκτιμήσουμε τις κοινέ αυτές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, τις κοινέ επιχειρήσεις, που είναι ο μοναδικός τελικά τρόπος που μας, επιτρέπουν, ε, που μας επιτρέπει να προωθήσουμε τα σημαντικότατα αυτά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να μιλήσω για την κοινή επιχείρηση Clean Sky. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την συνέχιση του προγράμματο αυτού. τρει παρατηρήσει Πρώτον, όσον αφορά την τροπολογία 13 και τον προπολογισμό. Με την τροπολογία αυτή μειώνεται ή προτείνεται μείωση περικοπή του προπολογισμού και θεωρώ ότι η προβλεπόμενη περικοπή θα μπορούσε ενδεχομένω να μειώσει τι θετικέ επιπτώσει τη κοινή αυτή επιχείρηση. Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ακόμα παρατηρήσει όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ε, η υφιστάμενη διακυβέρνηση στο πρόγραμμα Clean Sky 2 έχει δώσει θετικά αποτελέσματα. Βλέπουμε όμως ότι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αλλάξει κάπως τις ισορροπίες και ενδεχομένως να μειωθεί κάπως το σκέλος του ιδιωτικού τομέα. Ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό και να μην γίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερα, δεύτερον, όσον αφορά τις επιπρόσθετες δραστηριότητες, additional activities, Πρόκειται για συμπληρωματικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και εν μέρει ενδεχομένως από τον κρατικό τομέα. Πάλι εδώ πέρα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδεχομένως να απαιτήσει μια κάποια πολιτική δέσμευση προκειμένου να εφαρμοστεί. Και όσον αφορά την μόχλευση, το leverage, μιλήσαμε πάρα πολύ για το ζήτημα αυτό, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το ζήτημα της ε, δανειοδότησης. Σας ευχαριστούμε, Μάτσες Κουφόβιτς. Ε, Ευχαριστώ, Είναι σωστό ότι το ουσιαστικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ε, τι κάνουμε για να πρωτοπορήσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό τα προγράμματα ΣΔΙΤ είναι ένας μοχλός τον οποίο πρέπει να αναπτύξουμε, να πληροφορήσουμε ε, τους πολίτες μας, τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες ε, επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Πρέπει επίσης να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή της ορολογίας. Όταν λέμε κοινέ επιχειρήσεις και λέμε joint TISA, ε, δεν ξέρουν ακόμα και πολλοί ευρωβουλευτέ, περί τίνο πρόκειται. Τα ακρονίμια δηλαδή, ποιε είναι αυτές οι κοινέ επιχειρήσει, όποιο είναι εκτός του θέματος αυτού δεν έχει σαφή εικόνα. Είναι οι κοινέ επιχειρήσεις όπου συμπράττουν, ε, συμπράττει ο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ε, και οι πληροφορίες μας δεν πρέπει να διαδίδονται και να διανύμονται εδώ στις Βρυξέλλες αλλά και σε απόσταση 2.000 χιλιόμετρων. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτοί, αυτές οι πλατφόρμες να προσφέρουν πρόσβαση σε όλων των ειδών της επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσές, οι οποίες πλήττονται από την κρίση. αυτή η κρίση απέτησε την δημιουργία πολλών νέων πρωτοβουλειών ε, και καινοτομιών. Άρα αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι την πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων. Ευχαριστούμε κύριο Κορέγια Ντεκάμπος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να στηρίξω, να ευχαριστήσω και να στηρίξω το έργο του εισηγητή Παναγιωτόφ, του οποίου είμαι όδης ε, στη δικασία για τις ε, κυψέλες καυσίμου και την καύση τρογόνου να συμφωνήσω απολύτω με την μεγαλύτερη διαφάνεια από το περισσότερο ανοιχτό πνεύμα που χρειαζόμαστε. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση με την εμπιστευτικότητα, το απόρριτο. Η εμπιστευτικότητα έχει να κάνει με την ουσία. Η διαφάνεια με τη διαδικασία. Η διαδικασία πρέπει να είναι πλήρω διαφανή με πραγματική παρέμβαση του ε, Κοινοβουλίου στο peer review όπως προτείνεται από τον εισηγητή Παναγιώτο. Όμως πρέπει να αποσαφινιστούν και οι συνεισφορές σε ε, χρήμα ώστε να μην υπάρχουν ε, μικρές παρεκκλήσεις αλλά να δούμε και τι γίνεται με την ανακύκλωση των βασικών υλών, των απαραίτητων υλών ή τις νέες, τα νέα υλικά που απαιτούνται. Η συνένεσή μου λοιπόν εδώ είναι σαφής, ε, αλλά χρειαζόμαστε και σταθερότητα στον τομέα αυτό. Οι κοινέ αυτές επιχειρήσεις είναι μια καλή αφορμή για να έρθουν πιο κοντά η ακαδημαϊκή έρευνα με την επιχειρηματική ε, καινοτομία. Πάντως, η έμφαση αυτών των κοινών επιχειρήσεων δεν πρέπει να είναι επιπλέον ε, κονδύλια προς τον ιδιωτικό τομέα, αλλά ενίσχυση της εταιρικής σχέσης, της συνεργασίας, όχι υποκατάσταση λοιπόν. Να πω ότι η σημασία των ε, κεψελών καυσίμου. Σήμερα νομίζω ότι φάνηκε εύγλωτα και ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται να επιμείνω σε αυτό. Αλλά να πω ότι προχωρά ε, το θέμα αυτό παρά τον ανταγωνισμό της Κίνας και της Ιαπωνίας, οι οποίοι εργάζονται μάλιστα τάχιστα ως ανταγωνιστές μας. Γι' αυτό καλωσορίζω αυτήν την ε, προσπάθεια. Νομίζω ότι η έκθεση πάει στο σωστό, ε, στη σωστή κατεύθυνση και θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές στηρίζω τα συμπεράσματα του συναδέλφου Πανακετόφ. Ευχαριστώ τον κύριο Κορέγια Ντεκάμπους και τώρα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες στην συζήτηση αυτή, γιατί πρόκειται πραγματικά για ένα σημαντικότατο πακέτο επένδυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά αυτόν τον τρόπο συνολικά, δηλαδή σφαιρικά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Σας ευχαριστώ επίσης για τη σημασία που δώσετε σε κάποιες βασικές αρχές, το ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα των φύλων, διαφάνεια, προσβασιμότητα σε νέες αγορές, στο εμπόριο. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μία κλειστή λέσχη μια πολύ αρνητική εντύπωση που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο χρονικό διάστημα. Συμφωνούμε για τα αιτήματα τα οποία υποβάλλατε για απλούστευση, απλοποίηση, καθώς επίσης και για όλες τις υπόλοιπες παρατηρήσεις που κάνετε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα κάνω πρώτα κάποιες γενικές παρατηρήσεις και συνέχεια κάποιες πιο εξειδικευμένες. Όσον αφορά λοιπόν τι γενικέ παρατηρήσει, καταβάλουμε πολύ σημαντικέ προσπάθειε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλήξουμε στη δεύτερη γενιά των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών. Αντλούμε διδάγματα από τον πρώτο γύρο τέτοιων πρωτοβουλειών, προσπαθούμε τώρα να επιφέρουμε βελτιώσει, να εναρμονίσουμε τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούμε στα JTI, στι κοινέ τεχνολογικέ πρωτοβουλίε και να αποφύγουμε οποιαδήποτε επικάλυψη ανάμεσα στα κείμενα που έχουμε για τις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες, καθώς επίσης και τα γενικά κείμενα που έχουμε για τη συμμετοχή και για τις κατεξουσδότηση πράξεις, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα υπονομεύαμε την νομική ασφάλεια την οποία έχουμε πετύχει να αναφερθώ στο άρθρο 9, καθώς επίσης και στην διαδικασία απαλλαγής εκτέλεσης του προπολογισμού και θα αναφερθώ σε κάποια τεχνικά ζητήματα. Σας είπα ότι αντλήσαμε κάποια πρώτα διδάγματα από την πρώτη γενιά των κοινών επιχειρήσεων και όντως συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχε ένα υψηλότατο επίπεδο γραφειοκρατίας και ότι δεν μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να προωθήσουμε περισσότερο την εταιρική σχέση ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Έτσι λοιπόν αυτή τη φορά ακολουθούμε ένα νέο μοντέλο, το άρθρο 209, το οποίο όντως δίνει την απαραίτητη ευελιξία την οποία πρέπει να έχουμε για το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, για τη διαχείριση του προπολογισμού. Θεωρούμε λοιπόν ότι το νέο αυτό μοντέλο είναι πολύ καλύτερο. Πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτό το πρότυπο και γι' αυτό το λόγο βασιστήκαμε για τις βασικές διατάξεις σε αυτό το νέο άρθρο. Και αναφέρουμε εδώ πέρα και στο άρθρο 60 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, όπου προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την απαλλαγή, για την εκτέλεση προπολογισμού. Ξέρουμε ότι αυτό προκάλεσε κάποιους ε, δισταγμούς σε κάποιους συναδέλφους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε κάποιες άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά ουσιαστικά εκ των προτέρων εμεί θέλουμε να σας πούμε ότι κάναμε μία συζήτηση με τον βιομηχανικό κλάδο και τους διευθυντές των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι όντως υποστηρίζουν τη χρησιμοποίηση του άρθρου 209, συντοποιώντας ότι ε, αν επιστρέφαμε στο άρθρο 208 ως νομική βάση, το οποίο όπως σας είπα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό και ουσιαστικά αναφέρεται κυρίως στις, ε, στους ρυθμιστικούς οργανισμούς και όχι στις α, ε, συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα, τότε θα δημιουργούσαμε και περαιτέρω γραφειοκρατικό άκθος και περαιτέρω καθυστερήσεις. Και θα κινδυνεύουμε στην περίπτωση αυτή να μην τηρήσουμε τις ε, προθεσμίες μας και να μην ολοκληρωνόντουσαν κάποιες κοινέ επιχειρήσεις προτού προχωρήσουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές. Σας είπα λοιπόν ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω γραφειοκρατικό άχθος. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο αποφύγαμε να δημιουργήσουμε νέες συμβουλευτικές δομές. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες υποχρεώσεις υποβολής αναφορών πέρα από αυτές που υπάρχουν. Θέλουμε να διατηρήσουμε επίσης το επίπεδο προσωπικού χαμηλό και να έχουμε συγκεκριμένε και λίγες υποχρεώσει υποβολή αναφορά. Όσον αφορά τώρα τον προπολογισμό, σημαντικότατο ζήτημα. Ξέρετε ότι ε, η καινοτομία αποτελεί πλέον μία διάσταση στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε και να προασπίσουμε την καινοτομία. Να μην έχουμε απλώς ιδέες πρόθεσης κάποιων τεχνολογιών στην αγορά. Πρέπει λοιπόν ο ιδιωτικό φορέα να συμβάλλει περισσότερο και να επενδύσει περισσότερο στι κοινέ επιχειρήσει. Γι' αυτό τον λόγο θελήσαμε να εισάγουμε κάποιε επιπρόσθετε δραστηριότητε στα πλαίσια των συμπράξεων αυτών, των εταιρικών σχέσεων, πέρα από αυτά τα οποία προβλέπονται στο αρχικό τεχνολογικών πρωτοβουλειών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε τι νέε αυτέ δραστηριότητε με τη βοήθεια του ιδιωτικού φορέα. Συζητήσαμε επίση με το Συμβούλιο και συγκεκριμένα με την Κορεπέρ. Η στάση του είναι πολύ ενθαρρυντική, καθότι συμφωνούν με την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να μειωθεί ο προπολογισμό ή μάλλον προβλέπεται μια πολύ μικρή περικοπή για κάποιες κοινέ επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα για τα καινοτόμα φάρμακα. Όπως σας είπα, εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε μια οριζόντια περικοπή στο προπολογισμό, αλλά ενδεχομένως μόνο κάποιες επιμέρους διευθετήσεις. Ο κύριος Σέλερ, η κυρία Καβαγιό, η κυρία Αντρές Μπάρο αναφέρθηκαν στην δυνατότητα να έχουμε επιπλέον μεθοδολογικά μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν Όσον αφορά το διοικητικό κόστος, αυτό βρίσκεται στο 5%. Τώρα, για πιο συγκεκριμένες, κάποια πιο συγκεκριμένα σχόλια για κοινέ επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα κοινοτόμα φάρμακα, κάνουμε σημαντικές επενδύσεις γιατί πρέπει να ανταποκριθούμε σε πολύ σημαντικές κοινωνικές ανάγκες. Θέλουμε να κινηθούμε πιο επιθετικά προς την δημιουργία εξατομικευμένων φαρμάκων. Όσον αφορά το επιστημονικό πάνελ, συμφωνούμε ότι όντω θα πρέπει να συσταθεί. Είναι πολύ θετικό για διάφορε κοινέ επιχειρήσει, κοινοτόμα φάρμακα και άλλε. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση όμω να δημιουργήσουμε περιτέ επιπλέον συμβουλευτικέ υπηρεσίε. Ας εξασφαλίσουμε επίσης ότι ε, δεν θα δημιουργήσουμε ανάγκε επιτροπολογία, ακόμα και σε ομάδε εργασία που συμμετέχουν τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, πρέπει να σα πω ότι το χρονοδιάγραμμα εδώ συνάδει με το χρονοδιάγραμμα του Ορίζοντα 2020. Λάβαμε και την τελευταία πρόταση, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Όσον αφορά την κοινή επιχείρηση Excel, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοπορία. Σας διαβεβαιώ ότι θα, ότι θα έχουμε ελάχιστες αποκλήσεις και εξαιρέσεις προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα θέλαμε να είχαμε και μία αύξηση προπολογισμού για διοικητικούς κυρίως λόγους. Το είπε και ο κύριο Ρούμπικ αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προφανώ και εγώ και οι αδελφή, μου είμαστε στη διάθεσή για να απαντήσουμε σε τεχνικά ερωτήματα. Ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στους, διάφορες, στους διάφορους εισηγητές για μια τελική παρέμβαση, ο κύριος Οντή θέλει να επαναλάβει μια, ή να κάνει μια ερώτηση. Ναι, απλώς να επιστήσω την προσοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόβλημα τη ε, γραφειοκρατίας και τη απαλλαγή. Δεν είναι η διαδικασία τη απαλλαγή που προκαλεί γραφειοκρατικό άχθο. Η διαδικασία τη ε, απαλλαγή είναι μισή μέρα εκτελεστικών ε, διευθυντών που έρχονται να συζητήσουν με τους συζητητές και ένα δευτερόλεπτο ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο, καθώ και το ελεκτικό συνέδριο που έρχεται να ελέγξει όπω κάνουν όλοι οι ελεγκτέ. Αυτό προκαλεί γραφειοκρατικό άχθο και εδώ ήθελα την άποψη των εκτελεστικών διευθυντών, ιδίω των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν, είναι ότι αναγκάζονται να ευθυγραμμιστούν με τα δημόσια λογιστικά οι επιχειρήσει αυτέ. Αυτό είναι το τεράστιο γραφειοκρατικό άχθο. Έχουν τα δικά τους, το δικό του λογιστικό σύστημα, το ιδιωτικό, και εκεί ισχύει για αυτού το ίδιο σύστημα απαλλαγής. Καταλαβαίνω, Πατρίκο, ότι θα έπρεπε να είναι σαφέ όλο αυτό. Αλλά ένα δι για τι εταιρείε αυτές με λογιστική διαχείριση δημόσιου συστήματο νομίζω ότι είναι πολιτική αδεξιότητα. Θα πρέπει νομίζω λοιπόν να κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα για το θέμα αυτό. Ωραία. Για πέντε λεπτά ο λόγος στην κυρία Μαντουρέλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους μου τους συναδέλφους και την Κομισιόν για, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για τα σχόλια του. Εκτιμώ τα γενικά σχόλια, τα οποία σημείωσα προσεκτικά και τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις που αφορά την έκθεση καινοτομικών ε, φαρμα, φαρμακευτικών προϊόντων. Ο κύριος ε, Οντί ιδιαίτερα αναφέρθηκε ε, στην έκθεσή μου και τη σημείωσα όλες. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσω να ενσωματώσω όλες τις τροπολογίες. Ασφαλώς ορισμένες θα τις ενσωματώσω, ορισμένες θα πρέπει να συζητήσουμε πιο λεπτομερώς. Δύο γενικά σχόλια. Καταρχάς τις περικοπές ε, του προϋπολογισμού ε, όπου είναι αναγκαίες, αυτές προέκυψαν από τις άμεσες περικοπές του Συμβουλίου. Εμείς εξετάσαμε τους προϋπολογισμούς των ΣΔΙΤ, τις προτάσεις, τα κριτήρια της αριστείας και αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό των περικοπών μόνο σε απόλυτη ανάγκη. Μακάρι να μην είχαμε ανάγκη. Κύριε Οντή, όλοι θα προτιμούσαμε τα προγράμματα βάσει του άρθρου 187 να, να χρηματοδοτούνται και όχι βάσει του 186 τα κοινά προγράμματα δημόσιο-ιδιωτικού τομέα καλύπτονται και από το δικό του κανονισμό και εμείς ως εισηγητές θα προτιμούσαμε μια μεγαλύτερη συνέπεια. Ε, αυτά τώρα όλα αποτελούν μέρος της συμφωνίας και το Κοινοβούλιο οπωσδήποτε έχει έναν ε, μια καλύτερη συμμετοχή και ευθύνη ε, από ό,τι στο παρελθόν για τα ΣΔΙΤ βάσει των κανόνων ε, συμμετοχής που θα καλύπτονται από τις κατεξιοδότηση πράξεις. Άρα λοιπόν είμαστε σε κάπως καλύτερη μοίρα από την πρώτη γενιά των συμπράξεων δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Αυτά τα ΣΔΙΤ λοιπόν έχουν συζητηθεί ε, επιμακρών κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων και των συναντήσεων για τον ορίζοντα 2020. Επίσης έχουμε αρκετά, αρκετή εμπειρία από την πρώτη γενιά των συμπράξεων και θέλουμε να τροφοδοτήσουμε το αποτέλεσμα, τις συμπεράσματα αυτών των συζητήσεων στις αποφάσεις μας εδώ πιστεύουμε ότι έχουμε επιφέρει έναν ικανοποιητικό ρυθμό ε, συνοχής και συνέπειας με τον ορίζοντα 2020. Όπως σας είπα, θα διαβουλευθώ και με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για να προσπαθήσω να καταλήξουμε σε ένα γενικώ αποδεκτό συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Πρέπει αυτά τα, τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τα προγράμματα αυτά να τα εξετάσουμε ε, δηλαδή ε, το κάθε ξεχωριστά για να το αξιολογήσουμε και να δούμε κατά πόσο επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό ή όχι και αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα πρέπει να το εξετάσουμε ακόμα και ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που τονίστηκε τόσο πολύ από τους συναδέλφους η συμμετοχή του τομέα ε, η Ευρώπη έχει έχει σημειώσει τεράστια επιτεύγματα στον, ε, το, στους τομείς αυτούς, αλλά οι καινοτομίε, η έρευνα πολλές φορές δεν ε, υιοθετούνται από τον αρμόδιο τομέα, τον ιδιωτικό. Και λέμε πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί πρακτικά. Και πολλές φορές δεν γίνεται αυτά τα, τα διαμάντια των επιτευγμάτων παραμένουν χρησιμοποιείται. Πρόκειται για έργα για τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να ελοπιθούν. Πρέπει να επιβάλλουμε στην, στους ε, σχετικούς τομείς να συμμετάσχουν επιτέλους ε, να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους, τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, διότι όποιος δεν εξάγει εν τέλει δεν θα έχει και να φάει. Υπάρχουν και οι προτάσεις του συναδέλφου Ταλιάνη και ε, στο, το Μάρτιο ε, στο Συμβούλιο Κρατών και Αρχηγών, ε, Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων θα συζητηθούν αυτά τα θέματα. Ασφαλώς και η επικοινωνία και οι σαφείς ορισμοί παίζουν ένα ρόλο και πρέπει να είναι σαφείς. Στην Επιτροπή Περιφερειών ε, από την οποία προέρχομαι μιλήσαμε ε, μισή ώρα για αυτό το θέμα ε, σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δηλαδή του Κοινοβουλίου και οι, βιο... οι βιομηχανίες που βασίζονται στην βιοενέργεια παρουσιάζουν πάρα πολλές ευκαιρίες για τις περισσότερες περιφέρειες της Ένωσης και ιδίως τα καινούργια μέλη. Στα νέα μέλη η βιομηχανία χρησιμοποιείται περισσότερο και ωφελεί την Ήπεθρο και τις αγροτικές περιφέρειες. Δεν μιλούμε μόνο για τις κορυφαίες περιφέρειες, τις, τις καλύτερες, αλλά πρέπει να διαδοθούν οι βιοτεχνικές σε όλες τις περιφέρειες, ιδίως τις πιο αδύναμες συμφωνώ στη συζήτηση που έγινε με όλα τα θέματα ουσίας. Ο κύριος Έιλερ έχει το λόγο. Στο τέλος της ημέρας, τι θα κάνουμε. Υπάρχει η πρακτική πλευρά και η πολιτική πτυχή. Από τώρα, αν δούμε την πολιτική πτυχή, η Κομισιόν και το Συμβούλιο ας πούμε ότι δέχεται να τα, να τα χειριστεί όλα αυτά τις κοινέ επιχειρήσεις ως πακέτο. Χρειαζόμαστε κάποια ευελιξία από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Από πρακτικής απόψεως το πλεονέκτημα θα ήταν εάν κάνουμε καταρχάς τη διαβούλευση μετά τις πράξεις κατευθυνσιοδότηση μέσα σε μια δεδομένη σε δομή θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες έγκρισης του πακέτου. Εάν λοιπόν το κάνουμε όλο αυτό με έναν εμπεδομένο τρόπο, θα μπορέσουμε να βρούμε μια γρήγορη λύση. Και τώρα, πώς θα ε, εφαρμόσουμε την δομή συζήτησης, διαβούλευσης. Θα είναι ε, απλούστευση, ε, διακυβέρνηση και έτσι μπορούμε να δομήσουμε τη συζήτηση και με τους συγητές και με τα άλλα θεσμικά όργανα για το θέμα, το πρακτικό της απαλλαγής, για να είμαστε ειλικρινοί αυτή τα μία συμφωνία που έγινε μέσα στην, ε, στο χρηματοδοτικό κανονισμό. Ε, ξέρουμε ότι εάν ένα κομμάτι το αφαιρέσουμε, θα, θα υπόκειται στην απαλλαγή και στους συναφείς κανονισμούς. Μπορούμε όμως να αποσυνδέσουμε το θέμα ε, της απαλλαγής και να ε, εφαρμόσουμε πιο απλούς κανόνες, ε, αλλά παρόλα αυτά να υπόκειται στο πλαίσιο της εξωτερικής απαλλαγής. Δεύτερον, μέσα στα πλαίσια του προπολογισμού δεν νομίζουμε ότι εδώ ζητάμε μία προσωπική προσέγγιση κάθε εισηγητή όσον αφορά τις περικοπές. Πρέπει ιδίω για το, την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 πρέπει να σας πω ότι το όλο budget των μεταφορών υφίσταται ισχυρέ πιέσεις, περιοριστικέ πιέσεις διότι έχουμε το Clean Sky 2, έχουμε το Cesar, το Caesar πρόγραμμα και ε, τα άλλα επίπεδα 5 και 6 τα οποία είναι αρκετά κοντά στην αγορά. Υπάρχει συνεργατική έρευνα η οποία πρέπει να χρηματοδοτεί. Άρα λοιπόν σαφώς προκύπτει θέμα αναλογικότητος ε, στον προϋπολογισμό ε, ή δηλαδή από στρατηγικής απόψεως ίσως ε, θα θέλαμε να χρηματοδοτήσουμε πολύ περισσότερο το ένα καλά προγραμμάτων και όχι το άλλο. Αλλά από πλευράς ε, Κομισιόν δεν θα πρέπει να αποσυνδέσουμε ε, όλη αυτή την προσέγγιση πρέπει να είναι ισόρροπη και οριζόντια για να μην αντιμετωπίσουμε δυσκολίες αργότερα στις απαλλαγές των ε, κοινών επιχειρήσεων και των συμπράξεων, των ΖΙΤ. Πρέπει λοιπόν από τώρα να αναλογιστούμε το στοιχείο της αναλογικότητας ε, ε, των ε, μειώσεων και των απαλλαγών έτσι ώστε να μπορέσουμε να εγκριθεί όλο αυτό το πακέτο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις και πιστεύω πραγματικά ότι η Κομισιόν θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά δεδομένου ότι έχουν τα συμπεράσματα και έχουν, συνάγει και τα, ε, έχουν γνώσεις και εμπειρίες από την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση, την, την ενδιάμεση αξιολόγηση. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε μια συνάντηση συγητών και σκιωδών. Εγώ προσωπικά έκανα μια ενδιάμεση αξιολόγηση των ε, προγραμμάτων Τώρα ε, θα μπορούσε να προκύψει ένα πολιτικό πρόβλημα εάν μεμονωμένοι εισηγητές ε, προωθούν ή ασχολούνται μόνο με το τους ε, με τη δική τους κοινή επιχείρηση. Πρέπει, πιστεύω, όλοι οι συγητές να ακολουθήσουν μια κοινή γραμμή. Τα κοινέ αυτές επιχειρήσεις να διευθετηθούν σε ένα πακέτα πακέτο το Φεβρουάριο να κάνουμε μία εμπεδομένη συζήτηση για τις εξουσιοδότηση πράξης και να τελειώσουμε με το πακέτο μέχρι το τέλος Μαρτίου. Αλλά σε αυτή την ενιαία γραμμή. Ευχαριστούμε συνάδελφος Ρούμπι. <clears throat> Ευχαριστώ. Ε, πιστεύω ότι όλα αυτά που ήθελα να πω ελέγχθησαν. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την καλή συνεργασία. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια καλή δομή για να αυξήσουμε την αγορά απασχόλησης, τις θέσεις εργασίας ε, και το μέλλον της έρευνας και στην Ευρώπη. Ο κύριος Παναγιώτοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Тошновски, Брежина и Декампуш за отличните коментари, препоръки. Δεν έχουμε λοιπόν ε, καμία αντίρρηση στη γενική γραμμή. Ευχαριστώ όλους ε, τους συναδέλφους και την Κομισιόν για την υποστήριξη που μου έδωσαν. Ευχαριστώ και τον κύριο Βιτόριο Πρόντι, ο οποίος με βοήθησε ιδιαίτερα σε ένα κοινό, με μια κοινή εκδήλωση για το θέμα υδρογόνου και ανάπτυξη τεχνολογίας. Το οργανώσουμε μαζί αυτήν την εκδήλωση και ευχαριστώ και την Κομισιόν για την εμπεριστατωμένη της ανάλυση και για την επιβεβαίωσή της ότι προωθεί και εκείνη μια κοινή κατεύθυνση. Ο κύριος ε, Πρέχνερ μας, μου έδωσε καλές ε, υποδείξεις για την έκθεσή μου. Μου είπε ότι δεν υπάρχουν αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις που, που εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποίησης υδρογόνου, αυτού του καυσίμου και πιστεύω ότι θα καταρθώσουμε να ενσωματώσουμε τις νέες εξελίξεις στα προγράμματά μας, ξεπερνώντας τα προβλήματα. Πίστευω ότι η τεχνολογία των ε, κυψελών καυσίμων είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον ε, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση πράσινων καυσίμων. Θα ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν θέλει να απαντήσει, στην ερώτηση του συναδέλφου Οντί. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για το θέμα της απαλλαγής, θα ήταν όντως λογικό να γίνει συζήτηση για να βρεθεί κάποια λύση. Επιβεβαιώνω ότι έχουμε γραπτή βεβαίωση από τους ε, γενικούς διευθυντές των ε, κοινών επιχειρήσεων και του ιδιωτικού τομέα ότι συμφωνούν με το σχετικό άρθρο. η αρχή επιλογής, η αρχή για την απαλλαγή θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια, όμως εδώ είναι και η ουσία του ζητήματος. Δυστυχώς, οι δημοσιονομικοί κανονισμοί μας απαγορεύουν να γίνεται, να ε, εκτελείται απαλλαγή απευθεία για τις κοινέ επιχειρήσεις. Θα πρέπει να αναθερήσουμε τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό για το σκοπό αυτό, ε, κάτι που θα χρειάζεται καμιά διετία ή να παρεκκλίνουμε από τον δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό είναι κάτι που δεν πάω το προτείνω όπως φαντάζεστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε όμως προθυμότατοι να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα. Δεν είναι πραγματικά πρόβλημα, είναι κάτι που απλώς πρέπει να το βελτιώσουμε. Σας ευχαριστούμε. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για σήμερα το, τη συνεδρίαση για σήμερα το πρωί. Να θυμίσω ότι η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών είναι στην, την Τετάρτη στις 4 Δεκεμβρίου το μεσημέρι και να θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στις 15 η ώρα, στις 3, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση της Επιτροπής μας, όμως τις τέσσερις θα μιλήσουμε για το ίδιο θέμα, για το ΣΕΖΑΡ και τις υπόλοιπες κοινέ επιχειρήσεις. Σας ε, ευχαριστώ, θα το πούμε μετά.